Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε στην απογευματινή μας συνεδρίαση, όπου θα ακούσουμε μια παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Διαστημικών Προγραμμάτων που διευκολύνουν τις πολιτικές μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Πιέντερσο, τον Γενικό Διευθυντή και τον Διευθυντή Ματία Πέτσκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκτελεστικό διευθυντή Κάρλο Ντεστορίδη από τον οργανισμό GSA και την Πασκάλ Κλοντέλ που είναι από το GNSS και η κυρία Μάρτα Ψισόφσκα από τον Οργανισμό για το Ευρωπαϊκό GNSS, τον GSA. Η παρουσίαση θα καλύψει τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα που διευκολύνουν τις πολιτικές μας και που ενδιαφέρουν φυσικά και την Επιτροπή Ήτρε. Είχαμε την ε, νομοθετική έκθεση για το πολιτής δημοσιονομικό πλαίσιο του κ. Σαλίνη, το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα Γαλιλαίος και το GNSS, το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης ε, και το Κοπέρνικος στηρίζουν πολλές δραστηριότητες και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν την Επιτροπή Ήτρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν αποφασίσαμε να βάλουμε τα δυνατά μας και να καταλήξουμε συμφωνία για το διαστημικό πρόγραμμα πριν τις ευρωεκλογέ. Θα ακούσουμε μια παρουσίαση από τους καλεσμένους μας και θα ακολουθήσει συζήτηση μαζί τους. Παίρνω λοιπόν Αμέσω στο Πιέρ Show τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες επιχειρήσει. της DG Grow. Θα μα δώσει την προοπτική των διαστημικών προγραμμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγορά. Σα ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την συνάντηση και μα δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη διαστημική μα πολιτική. Κυρίω τη διαστημική πολιτική ω ε, μηχανισμό διευκόλυνση και άλλων πολιτικών. Χαίρομαι που είμαι εδώ, γιατί γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν θερμό υποστηρικτής των διαστημικών μα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών και, θέλω, και χρειαζόμαστε ακόμη την υποστήριξή σα και στο μέλλον, γιατί όπω είπατε η πρόταση για το ΠΔΛΤΑΠ δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχει εγκριθεί ακόμη επίσημα και θα θέλουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και τις συμφωνίες συνομοθετών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το διάστημα είναι σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας, παρόλο που μερικές φορές ε, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τη σημασία του. Και όταν ε, μιλάω στον κόσμο και τους λέω ότι συμμετέχω στην διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κόσμος με κοιτάει απορριμμένος και δεν ξέρει τι κάνουμε στο διάστημα και ποια είναι τα οικονομικά ωφέλη της διαστημικής πολιτικής και του διαστήματος. Γιατί ξέρουν ότι διάστημα είναι εκτόξευση δορυφόρου, μια δαπανηρή φυσικά πρωτοβουλία, αλλά δεν γνωρίζουν ότι σε μεγάλο βαθμό η καθημερινότητά του επηρεάζεται από το διάστημα. Γι' αυτό και είναι σημαντική η σημερινή συζήτηση και χαίρομαι ιδιαίτερω για την πρωτοβουλία σα να τη διοργανώσετε. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι είμαι πρόθυμο για συνέχιση διαλόγου και πέραν των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Θα πρέπει λοιπόν με το διάλογο που θα έχουμε να καταφέρουμε το διάστημα να γίνει προσιτό και στους Ευρωπαίους πολίτες και να αντιληφθούν πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Επίσης, το μήνυμά μου είναι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας στο διάστημα μέχρι στιγμής. Γιατί πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στα αρνητικά στοιχεία, στις αδυναμίες, στις αποτυχίες, στις δυσλειτουργίες. Αν εξετάσουμε όμως τα επιτεύγματά μας ε, ε, στη διαστημική πολιτική, είναι πολύ εντυπωσιακά. Το πρόγραμμα Κοπέρνικος, που είναι ένα σύστημα παρατήρηση, γεωπαρατήρησης άνευ προηγουμένου. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο ένα τέτοιο σύστημα. Το Κοπέρνικους προσφέρει άριθμα στοιχεία για τη Γη που χρησιμοποιούνται σε πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Ε, παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, της θάλασσας, ε, παρακολούθηση περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης. Το Κοπέρνικος λοιπόν είναι ένα εργαλείο απαράμιλο και άνευ προηγουμένου στον κόσμο. Και νομίζω ότι έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και όταν πρόσφατα οι Ηνωμένε Πολίτες αντιμετώπισαν τυφώνες και κυκλώνες, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουν τον Κοπέρνικο για να παρακολουθήσουν την κατάσταση στη Φλόριντα. Δεν έχουν κάτι αντίστοιχο. Οπότε μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το Κοπέρνικο. Και για το Γαλιλαίο το ίδιο. Ξέρω, είχαμε κάποια συμβάντα, είχαμε το blackout, είχαμε μια βλάβη. Αλλά αυτό που πετύχαμε με το Γαλιλαίο είναι ένα σύστημα που είναι σχεδόν λειτουργικό πια. Και ήδη δίνει υψηλή ποιότητα αποτελέσματα. Και δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί μόνο από ένα κράτος μέλος. Το Κοπέρνικους, το Γαλιλαίος και το Έγνος είναι παραδείγματα τη προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί χωρί την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα κράτο μέλο από μόνο του δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει τόσο μεγάλα επίβολα προγράμματα. Και καλό είναι να νιώθουμε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μα. Άλλο υπερήφανοι βέβαια και άλλο συγκαταβατικοί. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαυόμαστε στι δάφνε μα και να μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Υπάρχει και το μέλλον. Και γι' αυτό η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πιδελταπή είναι σημαντική, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε να οδεύουμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Και το τρίτο μήνυμα που θα ήθελα να σα μεταφέρω, μην φοβάστε, δεν έχω τόσα πολλά, θα είμαι σχετικά λακωνικός. Το τρίτο μήνυμα λοιπόν που θα ήθελα να σας μεταφέρω είναι ότι παρόλο που μερικές φορές δεν γίνεται αντιληπτό, θα πρέπει να φέρουμε το διάστημα στη γη. Δηλαδή να μεριμνήσουμε ώστε το διάστημα να γίνει εργαλείο που θα χρησιμοποιείται ακόμη περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και σε άλλους τομείς και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Γιατί μπορούμε από το διάστημα να λάβουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα βρούμε πουθενά άλλου. Οι συνάδελφοι θα σας δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε όχι μόνο για την Ευρώπη. Για παράδειγμα, αν θέλουμε για να παρατηρήσουμε κάτι στην Αφρική, οι εικόνες από το Κοπέρνικο θα είναι πολύ χρήσιμες για τον κόσμο εκεί, για τη γεωργία στην Αφρική. Με βάση τις εικόνες που δίνει το Κοπέρνικος και το Γαλιλαίος είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. θα σας τα εξηγήσουν οι συνάδελφοι εδώ. Πάντως είναι βέβαιο ότι ήδη το διάστημα είναι τμήμα της καθημερινότητάς μας. Παρόλο που μερικοί δεν το γνωρίζουν, δεν ξέρουν τι σήμα υπάρχει στο κινητό τους, δεν ξέρουν ότι όταν, όταν, όταν κάνουν ανάληψη ε, χρημάτων από τις τράπεζες, χρησιμοποιείται, χρησιμοποιούνται συστήματα IT από το διάστημα, δεν ξέρουν οι γεωργοί ότι όταν ψεκάζουν χρησιμοποιούν διαστημική τεχνολογία. Δεν το ξέρουν, αλλά είναι ήδη τμήμα της πραγματικότητας. Και τις προάλλες είχα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπήρχε μια συσκευή, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, ξεχωριστή και γκρίνιαξα κάπως γιατί δεν φαίνονταν και πολύ αποτελεσματικό το σύστημα και κάλεσαν έναν εμπειρογνώμονα και μου είπε όχι, αυτό το σύστημα είναι το καλύτερο που έχουμε γιατί λειτουργεί δορυφορικά παρόλο που δεν είναι μέσα στο, ενσωματωμένο στο όχημα. Και τα άλλα τι κάνουν, τα άλλα δεν ξέρω. Και αυτό είναι πραγματικά μια αληθινή ιστορία. Το διάστημα είναι μέσα στη ζωή μας πια. Και για να σας πω για το Κοπέρνικος, γιατί άλλοι θα μιλήσουν για το Γαλιλαίο, από τις εικόνες που λαμβάνουμε από το Κοπέρνικος, καταρχήν είναι τεράστιο ο αριθμό των εικόνων, εντυπωσιακό. Και ο Κοπέρνικος είναι από του μεγαλύτερου παραγωγού δεδομένων παγκοσμίω. Η πρόκληση όμω για μα είναι αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν για να καλύψει τις ανάγκες των ε, συμπολιτών μας, των επιχειρήσεών μας παντού. Και έχουμε ως καθήκον, και έχουμε καθήκον ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσουμε αυτά τα μαζικά δεδομένα να μπορούν να είναι εύχρηστα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε με τη δημιουργία ηλεκτρονικών πλατφορμών Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εικόνες που λαμβάνουμε από το Κοπέρνικους και υπάρχουν και εργαλεία για την επεξεργασία τους. Οπότε είστε μια μέρα στις Βρυξέλλες και βρέχει, μπορείτε να πάτε σε αυτήν την ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί από το κοπέρνικος για να αναπτύξετε νέες εφαρμογές, υπηρεσίες κτλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος. Έτσι φέρνουμε το διάστημα στη γη και αξιοποιούμε πραγματικά τα δεδομένα που λαμβάνουμε από το διάστημα. Και τέλος, κάτι που ελπίζω να υπάρχει στο νέο κανονισμό, είναι σημαντικό να έχουμε ένα ενιαίο μηχανισμό για όλα τα διαστημικά μας προγράμματα. Γιατί αυτό που θα χρειαστούμε στο μέλλον είναι οι συνέργειες στις εφαρμογές, στις υπηρεσίες, συνέργεια μεταξύ του Κοπέρνικο και του του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου. Αυτό χρειαζόμαστε. Θέλουμε συνδυασμό των υπηρεσιών και για τα ψηφιακά και για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και για την παρακολούθηση των μεταφορών. Θέλουμε να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τον Κοπέρνικο και α, από το Γαλιλαίο, από το γεω, γεωεντοπισμό του Γαλιλαίου. Και στο μέλλον θα μιλήσουμε για το ίντερνετ των πραγμάτων. Εκεί ο γεωεντοπισμός θα έχει μεγάλη σημασία. Και γι' αυτό η ποιότητα του Γαλιλαίου θα έχει τεράστια σημασία. Οπότε το συμπέρασμά μου θα ήταν ότι το διάστημα μετράει και δεν είναι κόστος, δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση. Γιατί όταν κατασκευάζεται κάπου μια γέφυρα, είναι δαπανήρη διαδικασία. Αλλά από τη στιγμή που διευκολύνει την κυκλοφορία, που ενώνει το Α με το Β σημείο, που διευκολύνει τη διακίνηση ανθρώπων, τη μεταφορά εμπορευμάτων, τότε η γέφυρα δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση. Το ίδιο και το διάστημα. Είναι επένδυση, όχι κόστος. Και το θέμα δεν είναι αν θα χρειαστούμε το διάστημα στο μέλλον. Φυσικά και θα το χρειαστούμε. Η ερώτηση είναι, θέλουμε την Ευρώπη να παραμείνει σημαντικός παράγοντας παγκοσμίω στα διαστημικά ζητήματα. Αυτό είναι το, το θέμα. Γιατί και η Κίνα κάνει μαζικές επενδύσεις στο διάστημα. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, υιοθετούν τη νέα προσέγγιση του διαστήματος, που ουσιαστικά προσελκύει ιδιωτικά κεφάλαια, τεράστια ποσά ιδιωτικά, που επενδύονται στον στο διάστημα, στον κλάδο του διαστήματο. Και δεν νομίζω ότι οι ιδιωτικοί επενδυτέ επενδύουν τα χρήματά του αστρονομικά ποσά γιατί του αρέσει το διάστημα, αλλά γιατί βλέπουν κέρδο από εκεί. Οπότε, ερωτώ, θα μείνουμε και εμεί στην κούρσα αυτή του διαστήματο ω Ευρώπη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η συμφωνία που ε, βρήκαμε για, την, ε, για τον κανονισμό MFF είναι σημαντική και είναι σημαντικό να διατηρηθεί χρηματοδότηση των διαστημικών προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ειλικρινά σας λέω ότι θέλω να συνεχίσουμε το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είμαστε στο ίδιο καράβι, έχουμε κοινό συμφέρον και είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση όποτε το επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να ε, κάλεσε τον κύριο Κάρλος Δεδορίζης που είναι επικεφαλής του οργανισμού ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Πλοήγησης του GSA και αν θέλουμε να μας δώσει τη δική του προοπτική για το διάστημα όσον αφορά τη βιομηχανία, τις αγορές. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε τρία, τρεις βασικούς στόχους. Το πρώτο είναι η συνεργασία και η παροχή υπηρεσίας. Η δεύτερη είναι η ασφάλεια. Και η τρίτη είναι η αγορά και η ανάπτυξη. Και δεδομένου του σημερινού θέματος θα εστιάσω σε αυτό το τρίτο άξονα. Τι, να, τι σημαίνει ακριβώς ε, αγορά ε, και ε, μάλλον επιρροή στην αγορά, θα σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα και θα ήθελα να ξεκινήσω με το άγνωστο που είναι ο προκάτοχος του Γαλιλαίου, ο πρόδρομος του Γαλιλαίου δεν είναι πολύ γνωστό κάθε φορά γιατί εμείς ως GSA ξεκινάμε από εκείνη την εμπειρία. Το άγνωστο λοιπόν είναι ένα σύστημα αύξησης που αυξάνει και ε, ενδυναμώνει το GPS σήμερα και τον Καλλιλέο αύριο και είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα όπου η υπηρεσία έχει αποκαλυφθεί στην κοινωνία της πολιτικής αεροπορίας τον Απρίλιο του 2007. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Να πω ότι αυτή τη στιγμή τότε ε, το έγνωση ήταν το πρώτο πανευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης. Δεν υπήρχε κανένα άλλο τέτοιο σύστημα. Άρα λοιπόν το θέμα ήταν ποιος θα πιστοποιήσει αυτό το σύστημα για την ε, πολιτική αεροπορία. Κανείς ε, δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να το κάνει αυτό. Και πώς θα κατανεμηθούν οι ευθύνες ανάμεσα στους διάφορους φορείς όσον αφορά ας πούμε τους προμηθευτές ε, ε, ε, πολιτικής αεροπορίας, τους παρόχους του έγνος, τα, πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την ενημέρωση, το, την τεχνολογική της αβιονικής. Εμείς προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να βρούμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Σήμερα μπορούμε να δούμε λοιπόν ότι έχουμε 26.000 πτήσεις το μήνα που χρησιμοποιούν το έγνος. Έχουμε επιπλέον 350 αεροδρόμια τα οποία είναι εξοπλισμένα με το έγνος. Έχουμε πάνω από 50% των ε, ε, διαδρόμων προσγείωσης στην Ευρώπη που ε, γίνεται η διαδικασία προσέγγισης με βάση το έγνος. Το GSA ήταν ε, καθοριστικό στο να γίνουν όλα αυτά, να συνδεθούν μεταξύ τους οι διάφοροι φορείς, να φέρουν τις προτάσεις τους και εδώ έχουμε τα αποτελέσματα. Και τώρα παραθέτω την πολιτική αεροπορία, γιατί το έγνος έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για την πολιτική αεροπορία, αλλά θα μπορούσα επίσης να πω ότι το έγνος ξεπερνά πολύ τον τομέα αυτό. Ε, γιατί χρησιμοποιείται για την ακρίβεια στη γεωργία, στα διόδια, ε, στους, στον υπόγειο ε, και ούτω καθεξής. Δηλαδή χρησιμοποιείται κατά κόρονα. Ας επανέλθω στον Καλλιλέο, το οποίο έχει ανακοινωθεί ότι θα άρχιζε τις υπηρεσίες του το τέλη του 2016. Και πάλι το GSE εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να έχει τα αποτελέσματα, να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα, καταρχάς κατανοώντας την δυναμική της αγοράς. Ποιοι ήταν δηλαδή οι κύριοι φορείς στην αλυσίδα αξίας. Έχουμε Ποιον πιστεύουμε ότι έπαιζε καθοριστικό ρόλο για την ε, την αγορά και την ε, αποδοχή από την αγορά. Έχουμε συνεργαστεί με τους κατασκευαστές, έχουμε δοκιμάσει τα προϊόντα τους και αν σήμερα έχουμε να εντοπίσουμε ένα δις δέκτες που πολλούνται παγκοσμίω, αυτό ακριβώς προέρχεται από αυτή την απόφαση, δηλαδή να ξεκινήσουμε την αρχική υπηρεσία στα τέλη του 2016 αλλά κυρίως ε, συνδέεται, μάλλον προέρχεται από την ε, σύνδεση των αναγκών όλων αυτών των φορέων. Λιγότερο από τρία χρόνια αργότερα λοιπόν βλέπουμε αυτά τα τεράστια εντυπωσιακά νούμερα, αλλά αν δούμε άλλους τομεί όπως ε, και τα αυτοκίνητα ας πούμε, τα αυτοκίνητα άνευ θα δούμε ότι και εκεί αυξάνεται το ενδιαφέρον για τον Γαλιλαίο Όλοι συνεργάζονται μαζί μας για να, δοκιμάσουν τα νέα χαρακτηριστικά και τα νέες συσκευέ που θα αποτελέσουν τη βάση του αυτόματου ε, και άνευ οδηγού αυτοκίνητου. Να σας, σας είπα τι γίνεται τώρα και να σας πω ότι προβλέπετε με τον νέο κανονισμό που θα αρχίσει να ισχύει σε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό για το GSA γιατί ε, λόγω του περιμέτρου των ευθυνών που θα διευρυνθεί. Ιδιαίτερα θα πρέπει να εστιάσουμε στο ότι υπάρχει μια θετική σύμπτωση. Ο νέος κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει, θα τεθεί εν ισχύ πάνω κάτω με το που θα έχει φτάσει στην πλήρη του απόδοση τον Γαλιλαίο. Θα έχει δηλαδή πλήρως αναπτυχθεί και μετά οι πλήρες υπηρεσίες ε, του θα ανακοινωθούν ε, ε, στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε γι' αυτό το ορόσημο και, και μαζί εμείς και οι υπόλοιποι φορείς να ετοιμαστούμε για αυτή τη νέα φάση όπου θα εστιαστεί η προσοχή στην παροχή υπηρεσίας. Αυτός ήταν ένας πρώτος στόχος. Ο δεύτερος είναι οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη της αγοράς. Θεωρούμε πως πρέπει να αλλάξουμε την ταχύτητα και τον όγκο των επενδύσεων που πρέπει να κάνουμε για την ε, ε, αποδοχή από την αγορά αφού τώρα μπαίνουμε στην φάση ε, παροχής των υπηρεσιών και αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε διάφορες ιδέες που θα πρέπει να μας επιτρέψουν να έρθουμε για να έχουμε αποτελέσματα του Γκαλιλαίου που θα ε, ε, αφορούν όχι μόνο τον τομέα των μεταφορών αλλά ε, και όπως σας είπα τη γεωργία ακριβίας και όλες τις βασικές τεχνολογικές τάσεις. Γεω... Εντο... είναι η βάση για όλα αυτά. Αυτά έχω να σας πω και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πασκάλ Κλοντέ. Είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού GNSS. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τις διάφορες δραστηριότητες της ε, Ευρωπαϊκής Δορυφορικής Πλοήγησης. Το GSA είναι ο οργανισμός για το Ευρωπαϊκό GNSS, δηλαδή προσφέρει ε, τις υπηρεσίες του έγνος και το γολιλαίο, σύστημα εντοπισμού θέσης και δορυφορικής πλοήγησης και στηρίζεται σε μία σύνθετη υποδομή που έχει ένα τμήμα ε, διαστημικό και ένα σκέλος επίγειο. Το σκέλος του διαστήματος απαρτίζεται από γεωστατικούς δορυφόρους και, το, ε, και τους εκτοξευτήρες και το σύστημα του εδάφους, ε, το επίγειο, διαχειρίζεται το σύνολο και αποτελείται από κέντρο ελέγχου και κέρες. Το Γαλιλαίο στηρίζεται σε ένα περίπλοκο σύστημα και υποδομής. Προβλέπει μια, ένα συγχρονισμό δισεκα, σε ακρίβεια δισεκατομμυριωστού του δευτερολέπτου που δίνει πολύ ακριβείς υπηρεσίες ε, θέσεις και χρόνου. Και επίσης έχει μια στοιχεία 22 δορυφόρων, επιχειρησιακών δορυφόρων σε τροχιά. Ε, μάλιστα έχετε όλοι στα smartphone σας ε, τέτοιες υπηρεσίες. Επίσης έχουμε υπηρεσίες ε, έρευνας και διάσωσης που σε, μέσα σε 10 λεπτά επιτρέπει τον εντοπισμό κάποιου με ακρίβεια ενό χιλιόμετρου και επίσης έχουμε και τις κυβερνητικές υπηρεσίες για τις κυβερνητικές αποστολές. Ο Κάρλο μίλησε για το Έγνωστο. Το έγνος είναι μια περιφερειακή υπηρεσία που καλύπτει το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακρίβεια του είναι τη ε, τάξη του ενό μέτρου και είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται κυρίω από την πολιτική αεροπορία αλλά και από τη γεωργία. Ε, ο οργανισμό GSA δεν είναι μόνο ένα οργανισμό που εξυπηρετεί την πολιτική του διαστήματο αλλά και του χρήστε, πολιτικού, θεσμικού και κυβερνητικού ο ε, οργανισμός GSA έχει ως επίκεντρό το χρήστη και η ανάπτυξη της αγοράς των χρηστών είναι η δεύτερη μεγάλη επιβολή αποστολή του οργανισμού μας. Και μάλιστα αξιοποιούμε τα σήματα που λαμβάνουμε από το διάστημα για όλα τα τμήματα της αγοράς προκειμένου να βρούμε καινοτόμες λύσεις. Αυτές οι καινοτόμες λύσεις που αφορούν εφαρμογές και δέκτες ε, τονώνουν το σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κλασικούς ε, βιομηχανικού κλάδου. Έτσι, όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τέτοιων καινοτόμων λύσεων, γιατί δεν χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερε ικανότητε στο διάστημα. Και η οικονομική ανάπτυξη που προσφέρεται από τέτοιο σύστημα δορυφορική ε, πλοήγηση εξυπηρετεί το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα σήματα του διαστήματο βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο μια τεχνολογική επανάσταση και αποτελούν ένα ουσιώδη καταλήτη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και αυτό ονομάζουμε downstream, μεταγενέστερη αγορά ή κατάντη αγορά. Και γι' αυτό ο οργανισμός GSA βρίσκεται στο κέντρο της νέας διαστημικής πολιτικής Made in Europe, πέραν τη παραδοσιακή διαστημική πολιτική. Επίση έχουμε πλατφόρμες χρηστών. Εκεί συγκεντρώνουμε και ε, κάνω μια ανάλυση του συνόλου των, των αναγκών των ε, τομέων τη οικονομία, μεταφορέ, γεωργία, πολιτική προστασία, τράπεζα, ενέργεια, για να βρούμε τα κατάλληλα προϊόντα για τι αγορά. Και έτσι ο οργανισμός μας συγκεντρώνει στοιχεία και αποκτά σημαντικές γνώσεις για την αγορά, κάτι που μας επιτρέπει να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες 2021-2022, υψηλής ακρίβειας ε, της τάξης 20 εκατοστών, για να έχουμε αυτόνομα οχήματα. Επίσης, ε, ε, υπηρεσίες εξακρίβωση ταυτότητας ή την υπηρεσία χρονομέτρηση και συγχρονισμό για τις κρίσιμες υποδομές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και το ορίζον ε, Ευρώπη και τα στοιχειώδη στοιχεία για τον οργανισμό μας, γιατί έτσι θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και ο προπολογισμό των δύο αυτών μηχανισμών θα έχει κεφαλαιώδη σημασία για το σύνολο του επιχειρηματικού ιστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οργανισμό μα δίνει το παρόν και στα περιφερειακά κέντρα αριστείας, αναπτύσσει προϊόντα που ανταποκρίνονται τι ανάγκε και τι προτεραιότητες των χωρών και με την τεχνογνωσία μας, με την ε, ε, παροχή υπηρεσιών και την τεχνογνωσία μας μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Επίσης, η αγορά downstream συμβάλλει τα μάλα στην μετάβαση προς μια πιο έξυπνη κινητικότητα και οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Επίσης, με το Smart Cities έχουμε πιο αποτελεσματικές ε, υπηρεσίες ε, βελτιστοποίηση ενέργειας και μεταφορών και διαχείριση των απορριμμάτων. Επίσης, η δορυφορική πλοήγηση βελτιστοποιεί τις διαδρομές των οχημάτων, μειώνει τη χρήση καυσίμων και την χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Και μάλιστα η συμβολή της δορυφορικής πλοήγησης έχει και κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. 10% της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται από τις δορυφορικές υπηρεσίες και είναι το 1 τέταρτο του, της παγκόσμιας αγοράς του διαστημικού downstream. 50.000 θέσει εργασία δημιουργούνται και 60 δισεκατομμύρια είναι τα έσοδα στην Ευρώπη από το Γαλιλαίο και το Έγνος μέχρι το 2027. Οπότε, η τεχνογνωσία που συγκεντρώσαμε στον οργανισμό με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνδυασμό με τον νέο κανονισμό διανοίγουν μεγάλες προοπτικές για το βιομηχανικό ιστό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. μέσω συνεργίας ε, μεταξύ του Γαλιλαίου, του Έγνος, του Κοπέρνικου και του GovSatcom. Έτσι μπορούμε να συνδυάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα του διαστήματος για να βρούμε ε, αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις. Μόλις συμπληρώσαμε τα 15 χρόνια λειτουργία μας και νομίζω ότι έχουμε όλα τα του για να φέρουμε τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κορονίδα του κόσμου. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή σας, την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε για όλη την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στον οργανισμό μας, όπως φαίνεται και από τις αποφάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα... Ακούσουμε τον κύριο Ματίας, ε, τον επικεφαλής των δολοφορικών προγραμμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να συμπληρώσω τα όσα ήδη ακούστηκαν. Να τονίσω και πάλι την στρατηγική διάσταση των διαστημικών προγραμμάτων. Το βάρος ε, το οποίο ρίχνουμε εμείς ε, στις ανάγκες ε, του χρήστη που είναι πραγματικά ένας παράγοντας ο οποίος μας διαχωρίζει. Το δεύτερο σημαντικό το οποίο μας διαχωρίζει είναι οι ποικιλίε οποίες η ποικιλία των υπηρεσιών. Παρέχουμε ανοιχτή υπηρεσία, ρυθμιζόμενη υπηρεσία προς ε, τα κράτη ως μέρος του πακέτου αρχικών υπηρεσιών. Τώρα για να συμπληρώσω τα όσα είπαν, θα εστιάσω στον ρόλο της ε, Κομισιόν. Το τι κάνουμε, τη στενή μας ε, συνεργασία με την GSA προφανώς και στο ότι εμείς ε, δίνουμε βάρος στις δυνατότητες που μας δίνει το διάστημα γιατί όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχει ήδη αυτή η διάσταση με τους δορυφόρους, με τα σήματα, με τα δεδομένα του Κοπέρνικου και προφανώς ε, πρέπει να φροντίσουμε στην γη να χρησιμοποιούμε τον καλύτερο τρόπο αυτές τις υποδομές. Έχουμε τα λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου για αυτές τις υποδομές και πρέπει να φροντίσουμε πραγματικά να χρησιμοποιούνται σωστά και επικέρδως. Όταν μιλάμε για τα λεφτά πρέπει επίσης να γνωρίζουμε πως πέρα από το ότι ε, είναι ένα σημαντικός ε, παράγων ε, και βεβαίως τέθη αυτό και για τον ρόλο του νομοθέτη η ΕΠΑ η οποία έχει υψηλότερο έποπτο από ΗΠΑ συγκριτικά ξοδεύει λιγότερα στο διάστημα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό λοιπόν εξετάζοντας τώρα τον ρόλο της Κομισιόν στις διάφορες δραστηριότητες πρέπει και πάλι να γνωρίσουμε πως το διάστημα είναι παρόν στην ε, καθημερινή μας ζωή. Ξέρουμε πως υπάρχει κάτι στα κινητά μας, αλλά ξεχνάμε την, ότι η λειτουργία του δικτύου αυτού απαιτεί έναν συγχρονισμό ε, Οπότε χωρίς ε, δορυφορική πλοήγηση δεν θα υπάρχει δίκτυο τηλεφωνίας, όχι μόνο για τις υπηρεσίες ε, τοποθεσίας, αλλά για βασικές υπηρεσίες για τις λευκοινωνιακές εταιρείες. Σε παγκόσμια κλίμακα έχουμε τους αριθμούς για την Ευρώπη, έχουμε τεράστια εξάρτηση λοιπόν από την διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών. Ξέρουμε ότι 10% του ΑΕΠ μας εξαρτάται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από την διαθεσιμότητα δορυφορικής πλοήγησης. Λοιπόν, τι κάνουμε ως Κομισιόν. Κάνουμε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι να αναλάβουμε την αναγκαία δράση ειδικά για λόγους ασφαλείας, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο. Σχολούμαστε στον τομέα της τυποποίησης καθώς αυτή βοηθάει στην υιοθέτηση και προσπαθούμε να ε, προωθήσουμε καινοφανείς και νεοφυείς επιχειρήσεις. Βεβαίω, η ρυθμιστική διάσταση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε ζητήματα ασφάλειας. Παραδείγματος χάρη, κρίσιμες υποδομές. Γνωρίζουμε ότι, όπως ήδη ακούστηκε, βασιζόμαστε σε αρκετές κρίσιμες υποδομές όπου ο συγχρονισμός ε, των ε, σημάτων παίζει έναν ρόλο στα δίκτυα τηλεπικοινωνίας, ε, δίκτυα ηλεκτρισμού ή χρονική σφραγίδα στον τομέα των τραπεζών. Όλα αυτά εξαρτώνται αυτή τη στιγμή από την διαθεσιμότητα του GPS. Εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα του σήματος GPS. Οπότε θα συνεχιστεί αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Ένα άλλο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο έξυπνος ε, ψηφιακός ε, ταχογράφος. Έχουμε ήδη αναλάβει δράση εδώ και απαιτούμε μέσω ε, κανονισμού που εγκρίθηκε πριν από 2-3 χρόνια ότι από τον Ιούνιο του 2019 τα φορτηγά θα πρέπει να έχουν έξυπνο ταχογράφο συμβατό με τον Γαλιλαίο. Δεν σημαίνει όμως ότι καθιστούμε υποχρεωτικά ε, υποχρεωτικό μόνο τον Γαλιλαίο. Πάντα έχουμε μια λύση ε, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον Γαλιλαίο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης. Όχι αποκλειστικά. Ένα άλλο θέμα που αφορά την ασφάλεια, πολύ επίκαιρο, είναι η πρωτοβουλία 112 που ενέκρινε η Κομισιόν και βεβαίως θα εντοπίζεται η θέση του καλούντος στην περίπτωση ανάγκης και θα μεταδίδεται στις υπηρεσίες ανάγκης. Είναι δηλαδή σαν τον κανονισμό για τα αυτοκίνητα και βασικά μεταφέρουμε το μοντέλο αυτού του κανονισμού που ισχύει για το αυτοκίνητο και είναι πολύ βασικό κομμάτι της ασφαλείας των αυτοκινήτων στα κινητά τηλέφωνα και θα υπάρχει έτσι η δυνατότητα τα κινητά τηλέφωνα σε περίπτωση ανάγκης προφανώς να δίνουν το στίγμα ε, του ατόμου που καλεί. συγκεκριμένα παραδείγματα τώρα ρυθμιστικών δράσεων που αναλύθησαν το, στο παρελθόν ή έρχονται τώρα. Δεύτερο παράδειγμα. Ε, απλά να το αναφέρουμε είναι η τυποποίηση. Μέσω της τυποποίησης έχουμε την ευκαιρία να διασφαλίσουμε ότι το Γαλιλαίο και το έγνος θα είναι όσο το δυνατόν πιο σημαντικά για τις αγορές. Οι υποδομές που έχουμε θα είναι όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμες ε, στον πραγματικό κόσμο και αυτό οφείλεται σε διάφορες διαδικασίες τυποποίησης στα σχετικά φόρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι όταν μιλάμε για ασφάλεια θα φροντίσουμε το έγνωσο να είναι εκεί και να χρησιμοποιείται μέσω των προδιαγραφών που θα καθορίζονται. Το ίδιο και για τις οδικές μεταφορές. Και πιο συγκεκριμένα τα αυτόνομα οχήματα. Υπάρχουν διαφορές δραστηριότητες. Εκεί όπου τη βλέπουμε μαζί με τις ρυθμιστικές αρχές έτσι ώστε για το θέμα των αυτόνομων οχημάτων ο Γαλιλαίος να χρησιμοποιείται το ίντερνετ των πραγμάτων. Είναι το τρίτο θέμα. Δηλαδή θα πρέπει εδώ πέρα οι σχετικές προδιαγραφές να περιλαμβάνουν το Γαλιλαίο και το Έγνος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Ροστόφσκα. Κρυβάνης Μπροστόφσκα, επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης ε, στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Ε, Έχετε λοιπόν τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Η σημερινή μου ε, εισήγηση θα προσιλωθεί στην ε, αποδοχή και από την αγορά ε, του συστήματος EGNSS. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι πολύ καλά νέα. Πριν από μερικές εβδομάδες φτάσαμε ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Διαπιστώσαμε ότι έχουμε ένα δις χρήστες CGNSS και αυτός ο αριθμός των χρηστών αναπτύσσεται ακόμα, ε, αυξάνεται διαρκώς γιατί όπως μόλις ακούσατε το EGNSS είναι ένα σπουδαίος και βασικός μεσολαβητής για την ανάπτυξη διαφόρων άλλων τεχνολογιών. Αυτό ε, το σύστημα έχει ήδη γίνει δεκτό γιατί η βασική του λειτουργία είναι ένα διαμεσολαβητή Ήδη 600 ε, διαδικασίες ε, που βασίζονται στο έγκνος σε πάνω από 330 αεροδρόμια στην Ευρώπη. Επίσης, 83% ε, των νέων τρακτέρ είναι ήδη λειτουργούν, μπορούν να λειτουργήσουν με το EGNSS η οδηγία περί του νέου ταχυγράφου έδωσε νέα όθηση στην αγορά και χάρη σε αυτό υπάρχουν 17 μάρκες αυτοκινήτων που ε, βάζουν στην αγορά το Έγνος και το Γαλιλαίο. Αυτά είναι παραδείγματα, αλλά όλα αυτά τα νούμερα εύκολα μπορούν να μεταφραστούν στα ωφέλη ε, που αποκομίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν γέννη, λοιπόν, χάρη στο έγνος έχουμε πολλές ε, καθυστερήσεις οι οποίες έχουν ε, αποφευχθεί. 50.000 θέσει απασχόλησης ετησίω δημιουργούνται στην Ευρώπη χάρη στο GNSS. Ε, Βελτιώσεις δε στις μεταφορές και στην αποτελεσματικότητα αυτών σημαίνουν ότι εξοικονομούνται 3,5 δις λίτρα καυσίμων και ε, και 15 ε, εκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα εξοικονομούνται χάρη στις βελτιώσεις αυτές. Αυτά όλα επιτυχάνονται λόγω της ολοκληρωμένης μας προσέγγισης όσον αφορά την ε, διείσδυση του, του EGNSS στην αγορά. Αφορά δε όλους τους τομείς της αγοράς, οι μεταφορές, ε, τις μαζικές αγορές, ε, εποπτεία γεωργική, ε, χρονισμός, συγχρονισμός και σε όλα αυτά τα, τα, τα μερίδια της αγοράς δουλεύουμε σε όλη την αξία, στην αλυσίδα αξίας. Δηλαδή έχουμε εφαρμογές, ε, ανα, σχεδιαστές εφαρμογών, πιστωτές και τελευταίως τους τελικούς χρήστες. Πρέπει καταρχά λοιπόν να γνωρίζουμε την αγορά και την τεχνολογία και εδώ οι χρήστε βρίσκονται στο επίκεντρο. Μιλάμε στου ενδιαφερόμενου φορεί, διοργανώνουμε σεμινάρια, διαβουλεύσεις, ε, κάνουμε μελέτες ε, ικανοποίησης. Ένα παράδειγμα είναι το project που ξεκινήσαμε και ονομάζεται Stay Close to Member States και με αυτό την έρευνα εξετάζουμε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες τους ε, για να τους στηρίξουμε στην υιοθέτηση και στη χρήση του GNSS. Το, το συζητάμε επίση σε περιφερειακό επίπεδο και προσπαθούμε να του βοηθήσουμε να καταλάβουν τι ερευνητικέ και αναπτυξιακές δυνατότητε. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορέσει να παγιωθεί το GNSS στην αγορά. Αφού λοιπόν συγκεντρώνουμε όλες αυτές τις γνώσεις από τους ενδιαφερόμενους όλους ε, και τα συνδυάζουμε στην έκθεση Market and Technology, αγορά και τεχνολογία. Ή μάλιστα αυτή δημοσιεύεται τακτικά και θα υπάρχει σε λίγες μέρες στο διαδίκτυο, στο site μας, η τελευταία της εκδοχή. Αφού λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει όλες αυτές τις γνώσεις, θα πρέπει να κατανοήσουμε και την πλευρά της ζήτησης. Συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν για να στηρίξουμε την τεχνική πτυχή ε, όταν ορίζονται οι κανονισμοί. Συζητάμε με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς για να δημιουργήσουμε οδικούς χάρτες ε, που θα οδηγήσουν στην, στην υιοθέτηση του GNSS γνωρίζοντας την αγορά, γνωρίζοντας την τεχνολογία, καθώς και γνωρίζοντας τι ζητάει η αγορά, δημιουργούμε την προσφορά, επενδύουμε. Γιατί θέλουμε να έχουμε ε, ευρωπαϊκά προϊόντα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Horizon 2020 είναι αυτό που στηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή του GNSS, αλλά και τα θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν τα τους ε, πόμπους και τους δέκτες. Το πρόγραμμα Horizon 2020 ε, συνεχίζεται. Ε, θέλουμε να μπορέσουμε να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την μεθοδολογία που αφορά το Genesis και έχει αποδείξει την αξία της και σε άλλους τομείς. Βλέπουμε το Κοπέρνικους και ας πούμε και πολλά άλλα προγράμματα μεταξύ των οποίων πιστεύουμε θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ε, συνεργασία όπως το GovSatcom. Όταν χρησιμοποιούμε τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορούμε να στηρίξουμε τις εταιρείες για, εξαγωγή και, για εξαγωγές και να πιέσουμε και να οθήσουμε την ε, αποδοχή από την αγορά. Για να ακόμα πιο ανταγωνιστικό ε, η ε, ε, ανταγωνιστική Ευρώπη στον διάστημα, θα πρέπει να ξεκινήσουν και άλλες πρωτοβουλίες. Δημιουργία εγχώριας αγοράς για τον Καλλιλέο, που θα συμμετέχουν περισσότερο οι δημόσιες αρχές όταν, όσον αφορά την υιοθέτηση του GNSS και να στηρίξουμε βέβαια τις μικρομεσαίες και τις ε, ε, νέες εταιρείες, τις startups. Δουλεύουμε λοιπόν σήμερα για την ε, αποδοχή από την αγορά και αύριο μεθαύριο χάρη στι νέες πρωτοβουλίες και τομεί. θα πρέπει να αναπτυχθούμε, να έχουμε νέα εργαλεία. Στόχος είναι το Γαλιλαίο να αποτελέσει το πρώτο από όλους ανάμεσα στους διάφορους ανταγωνιστές ώστε να επιφέρει να σημάνει τη διαφορά ε, Πολύ σημαντικό είναι επίσης να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς στις GNSS που είναι τώρα το 25%. Θέλουμε να το, να, να το αυξήσουμε τουλάχιστον στο 33% όπως και σε άλλους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Με τα χαρά λοιπόν να συζητούμε μαζί σας τα θέματα αυτά και σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Very Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε όλους για τις παρουσιάσεις που μας κάνατε. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τον κύριο Σαλίνη που ήταν ε, ο εισηγητής της Ήτρε για το διαστημικό πρόγραμμα. Έχετε το λόγο κύριε Σαλίνη. Σας ευχαριστώ. Εγώ ως πολιτικός είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την τεράστια πρόοδο που έχουμε σημειώσει στο διαστημικό πρόγραμμα. Και ως εισηγητής για το διαστημικό πρόγραμμα θεωρώ ότι η προσέγγιση μας στις διαπραγματεύσεις είναι σωστή και συγκεκριμένη και άρτια και επίση έχει, έχει μακροπρόθεσμη προοπτική. Και μάλιστα είμαστε και κάπως οραματιστές στις διαπραγματεύσεις. ονειροπόλοι Ελπίζω αυτό αυτόν τον ενθουσιασμό και τον οραματισμό να τον διατηρήσουμε και στις νέες διαπραγματεύσεις του προπολογισμού, αποφεύγοντα το ταραχώδες τελευταίο τμήμα του τριμερούς διαλόγου. Γνωρίζουν οι συνάδελφοι περί τίνος πρόκειται. Πάντως το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερος αξιόλογο και μας ικανοποιεί. Επανέρχομαι τώρα στα θέματα διακυβέρνησης και προϋπολογισμού, αλλά πρώτα να τονίσω ένα άλλο θέμα. Έχω εντυπωσιαστεί τα μάλα από τον τεράστιο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασπάστηκαν αυτές τις προκλήσεις. Μιλήσαμε για την κατάντη αγορά, την downstream αγορά, τη μεταγενέστερη αγορά και νομίζω ότι και upstream και ανάντι είμαστε ταγοί. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς τώρα και με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουμε να προωθήσουμε και την κατάντη αγορά. Ξέρουμε ποιος είναι ο βιομηχανικός αντίκτυπος από τα στοιχεία που μας δώσετε. Για την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, για παράδειγμα, για την έξυπνη κινητικότητα, την ψηφιακή οικονομία, πολύ θετικά τα πλεονεκτήματα, πολλά τα πλεονεκτήματα. Και να δούμε πώς θα προωθήσουμε την ανάπτυξη αυτής της δευτερογενούς αγοράς, της downstream αγοράς Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει αρκετά. Έχουμε τεράστιο αριθμό για παράδειγμα, για τη δωρεάν χρήση της τεχνολογίας και θα πρέπει αυτή η κατάσταση να την τροποποιήσουμε και να την βελτιώσουμε. Ο πραγματικός αντίκτυπος της καταπληκτικής αυτής τεχνολογίας είναι τεράστιος. Και εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε όχι μόνο ποια θα είναι η σχέση μεταξύ των οργανισμών, αλλά πώς με τον προϋπολογισμό μας θα προωθήσουμε τέτοιο είδος προσέγγιση, αξιοποίηση όλων αυτών των επιτευγμάτων και στην αγορά και οικονομικά. Και επίση θα πρέπει να συνδυάσουμε τις αρμοδιότητες και τις ικανότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής όχι στα βιομηχανικά μόνο θέματα, αλλά κυρίως στη βιομηχανία. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες και τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα βιομηχανικά θέματα. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η βασικότερη πρόκληση. Ευχαριστούμε κύριε Σαλίνη. Οι άλλοι σκιώδεις ηγητές τώρα έχουν το λόγο. Ο κύριος Σογίνιο είναι ο πρώτος στο κατάλογό μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω πορτογαλικά, οπότε θα χρειαστείτε τη διερμηνία. Θα σε, ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για τις ε, διεξοδικές πληροφορίες που μας δώσατε για τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει τώρα να συμπληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο για να καταστήσουμε δυνατά και βιώσιμα όλα αυτά τα επιτεύγματα που μας παρουσιάσατε και να υλοποιήσουμε όλη αυτή τη φιλοδοξία ε, που μας ε, μετέφερε η ομάδα του οργανισμού GSA, του Οργανισμού Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού GNSS. Όπως είπε και ο εισηγητής μας, βρισκόμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία ή πολύ κοντά στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, αν και έχουν μείνει κάποιες εκκρεμότητες. Η χρηματοδότηση, για παράδειγμα. Οι σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Και κάτι άλλο που δεν είμαστε ακόμη σε θέση να προσεγγίσουμε, γιατί μας, μας λείπει μια σημαντική μεταβλητή και είναι ο αντίκτυπος του Brexit στο πρόγραμμα αυτό, αν και όταν λάβει χώρα το Brexit. Οπότε μπορούμε προς το παρόν να επικεντρωθούμε σε κάποια πιο γενικά θέματα. Πρώτον, χρηματοδότηση. Προτινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση αρκεί για να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα της φιλοδοξίας. 33% μερίδια αγοράς, όπως είπατε, για το GNSS. Επίσης, τι εταιρικές σχέσεις θα μπορούσαμε να έχουμε με τις κυβερνήσεις ή με τους τελικούς χρήστες ώστε να καταστήσουμε πιο εύρωστο οικονομικά το πρόγραμμα και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί απέναντι σε άλλες ε, μεγάλες δυνάμεις που είναι οι ανταγωνιστές μας στην παγκόσμια αγορά. Οπότε θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο ε, θα ενισχύσουμε το πρόγραμμα. Και σίγουρα όλα αυτά τα προγράμματα είναι σημαντικά για να υλοποιήσουμε και το φιλοπεριβαλλοντικό μας πρόγραμμα για να απαλλάξουμε την οικονομία μας από τον άνθρακα, για να υλοποιήσουμε τις έξυπνες πόλεις, την έξυπνη κινητικότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναδείξουμε αυτή τη διάσταση και να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας, να την προβάλλουμε καλύτερα, για να γίνει αντιληπτή από τους Ευρωπαίους πολίτες. Και πολύ συχνά ο απλός πολίτης σκέφτεται το διάστημα Ω κάτι που έχει σχέση με τον πόλεμο των άστρων, για παράδειγμα, ή ένα θέμα που αφορά κυρίω την άμυνα. Δεν σκέφτεται τι άμεσε συνέπειε που έχει στην καθημερινότητά του, στο επίπεδο τη ζωή του, στην, στο καθαρό περιβάλλον, στην απαλλαγή από τον άνθρακα. Τι τεράστιες υπηρεσίε προσφέρει το διάστημα στην ανθρωπότητα. Δεν το σκέφτεται αυτό ο θα πρέπει να το ενημερώσουμε. Σε ό,τι αφορά τι ε, τρίτε χώρε, ήμουν και ο για το ψηφιακό πρόγραμμα τη Ευρώπη και προσθέσαμε ένα άρθρο για τον διοντολογικό κώδικα που θα πρέπει να εφαρμοστεί στη σχέση με τις τρίτες χώρες. Τέτοια προγράμματα επηρεάζουν ιδιαίτερο τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές μας σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Εσείς πώς το βλέπετε. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα είδος ε, δεοντολογικής πιστοποίησης ε, στη σχέση μας με τις τρίτες χώρες για τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ κύριο Γκρουτιλέρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως και ο δισηγητής του διαστημικού προγράμματος έχω και εγώ κάποιες συγκεκριμένες απορίες. Κύριε Δελσό, οι Αμερικανοί εδώ και πολύ καιρό έχουν υιοθετήσει το νομοσχέδιο αγορά στα Αμερικανικά, Buy American, που επιβάλλει την αγορά Αμερικανικών προϊόντων στην Αμερικανική επικράτεια για τις άμεσες αγορές της Αμερικανικής κυβέρνησης, για τις κρατικές προμήθειες δηλαδή. Δεν κρίνεται σκόπιμο για να προστατεύσουμε εμείς το διαστημικό μας κλάδο να έχουμε κάτι αντίστοιχο. Για να έχουμε και έσοδα, όχι μόνο έξοδα. Μήπως θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ ενός Buy European Act, ενός ειδικού νόμου αγοράστε ευρωπαϊκά, τουλάχιστον για τον διαστημικό κλάδο. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους πόρους σας, και τους οικονομικούς και τους ανθρώπινους, έχετε τους απαραίτητου πόρου για να ανταπεξέλθετε στα σημερινά και τα μελλοντικά σας καθήκοντα και τι αποστολέ. Από ό,τι ξέρω έχετε 200 μόνιμους και συμβασιούχου. Σε σχέση όμως με το μελλοντικό κανονισμό για το διάστημα που σας επιφορτίζει με νέες ευθύνες, έχετε αρκετούς πόρου δημοσιονομικούς και ανθρώπινο δυναμικό για να ανταπεξέλθετε. Επίσης, εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τον οργανισμό GSA και θα ήθελα πολύ να λειτουργήσει εύρυθμα. Και ο οργανισμός και όλα τα σημεία της διαστημικής πολιτικής. Βλέπω στον κανονισμό για το διάστημα ότι όλα είναι προσδιορισμένα και η μελλοντική διακυβέρνηση επίσης είναι σαφώς οριοθετημένη. Όλα τα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο ασχολείται με την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και ο οργανισμό GSA ασχολείται με την ε, απόλυτη και αποκλειστική αξιοποίηση εκμετάλλευση των συστημάτων. Όλα αυτά είναι οριοθετημένα και πιστεύω ότι θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σωστά και να σημειώσουμε πρόοδο. Δεν ξέρω αν ε, δεν σας κατάλαβα καλά. Όταν μιλήσατε για το έγνος, είπατε ότι ο οργανισμός GSA θα ασχοληθεί με την ε, ανάπτυξη των συστημάτων. Ο κανονισμός όμως για το διάστημα προβλέπει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ασχολείται με την ανάπτυξη των συστημάτων. Μήπως δεν σας κατάλαβα καλά. Και τώρα που έχουμε ένα πλαίσιο που οριοθετεί τις αρμοδιότητες, έχουμε γερά θεμέλια για να αναπτύξουμε το διαστημικό μας κλάδο. Και αυτό θα συμβεί αν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων φορέων, προκειμένου μέσω της διαστημικής μας πολιτικής να προωθήσουμε τα ευρωπαϊκά μας ιδεώδη. Σας ευχαριστώ κύριε Στοσενόφσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική παρουσίαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχω τώρα κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, πρώτα απ' όλα. ο ναι, κύριο Ντελσό. Η επιστολή της κυρίας Γκουλάρ λέει ότι θα υπάρξει μια νέα διεύθυνση διαστήματος. Η βιομηχανία είναι πάντα πολύ ευαίσθητη. εγώ δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα με αυτό όσον αφορά την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στο Γαλιλαίο, αλλά θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη και να μου πείτε τι ακριβώς θα κάνει αυτή η νέα γενική διεύθυνση. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, στο Κοινοβουλίο και στην Επιτροπή μας, εδώ και πολλά χρόνια μιλάμε για το πώς ε, μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ε, ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσει που γίνονται από την ε, υπηρεσία ε, συστημάτων ε, κατεύθυνσης και βεβαίως αυτό είναι ίσως κάτι το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει εδώ πέρα στον τριμερή διάλογο. Μετά, τον κύριο να τον ευχαριστήσω για αυτά τα οποία επέτυχε, γιατί θυμάμαι ότι πριν από λίγα χρόνια ήμασταν σε ένα διοκτήριο στην ε, Πράγα και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ε, πλέον για το τοπίο αυτό είναι γεμάτο ζωή. Είναι πλέον το κέντρο της αστυνικής έρευνας στην Ευρώπη. Σας βγάζω λοιπόν το καπέλο. όλα αυτά Μιλάμε για μια κρίσιμη περίοδο. Ήδη ο Γαλλίος έχει αρχίσει να λειτουργεί, οπότε όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα έτσι, της παιδικής ηλικίας, αυτό προκαλεί και σε μας προβλήματα. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, πάρα πολλά λεφτά δίνουμε, γιατί βλέπουμε ακριβώς πόσες προοπτικές έχει. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποιο ε, θα είναι αυτό το επόμενο βήμα. Λοιπόν, κύριε Κλοντέλ, θα συμφωνήσω μαζί σας ε, για τις εμπορικές ε, δραστηριότητες. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά Ινστιτούτα. και να εκμεταλλευτούμε και το πρόγραμμα του Ορίζοντα. Και συμφωνώ επίσης με αυτό το οποίο είπε και ο κ. Ντελσό στην αρχή. διότι ο κόσμος το θεωρεί δεδομένο. Πηγαίνω στα πανεπιστήμια, όλοι πιάνουν το κινητό τους εκεί, κοιτάνε. Ε, δεν βλέπουν όμως ποια είναι η διαφορά από το GPS. Ε, το θεωρούν ε, το ίδιο πράγμα, εντάξει. Έχουν γαλιλαίο όμως και δεν είναι ακριβώς το ίδιο και πρέπει να το καταλάβουν. Ούτε θέλουμε να ενοχλούμε τον κόσμο και να λέμε να βάλουμε μια ειδοποίηση στο κινητό, να του λέμε ξέρετε έχετε και Γαλιλαίο. Αλλά πώς θα το μάθουν. Πρέπει να το γνωρίζουν, να το μάθουν ότι υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε συνάδελφοι τώρα, αλλά έχουμε καθυστερήσει λίγο, οπότε σα παρακαλώ να είστε λίγο πιο συμμαζεμένοι. Κύριε Μπομπά. Μάλιστα, κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ για τις εισηγήσεις σας. Ε, τα βρήκα όλα αυτά πολύ συναρπαστικά την πρόοδο δηλαδή του διαστημικού μας προγράμματος και των ε, επιμέρους προγραμμάτων. Έχετε δίκιο και το είπατε και ορισμένοι συνάδελφοι το είπαν επίσης ότι το θέμα του διαστήματος είναι πολύ σημαντικό ενώ ταυτόχρονα δύσκολα καταλαβαίνει ο κόσμος το συμφέρον που θα μπορούσε να έχει από την ανάπτυξη, να αποκομίσει μάλλον τα κέρδη που μπορεί να αποκομίσει την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων. Αυτά όλα και η εξάπλωση του έγνωστα θα απαντήσει νομίζω σε αυτά τα θέματα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να δούμε και το ε, οικολογικό ζήτημα και τον επίγοντα του χαρακτήρα και μιλήσατε για το Κοπέρνικο πριν από λίγο και ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα έχετε την αίσθηση και την εντύπωση πως η χρηματοδότηση που δίνεται σήμερα σε αυτά τα προγράμματα αρκεί αν κανείς δει τις προκλήσεις οικολογικού ε, τύπου και έπειτα υπάρχουν άλλα προγράμματα που να προβλέπονται για τη βελτίωση της μας, ε, γνώσης μας περί του πλανήτη και της κατάστασής του. Έπειτα, αυτό που είπε και ο συνάδελφος ε, όσον αφορά την συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη, τους οργανισμούς που εσείς εκπροσωπείτε, Έχω την αμυδρά εντύπωση ότι για να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που ε, έχουμε ενώπιόν μας, θα πρέπει να υπάρχει σαφέστερη κατανομή των καθηκόντων ε, μεταξύ όλων των οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αρμο... Ε, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επικαλύψεις, αλλά και ε, ίσως και επικαλύψεις κονδυλίων. Σας ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνεται ο γύρος των σκιωδών εισηγητών και έχω άλλους τρεις συναδέλφους που θέλουν να πάρουν τον λόγο. Παρακαλώ όμως να περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τους ομιλητές για τις ε, παρουσιάσεις. Όλο το πρωί ήμουνα σε μια συνεδρίαση για το Brexit και ε, επιτέλους χάρηκα που ήρθα εδώ από μια αρνητική κατάσταση, εντελώς αρνητική. Χαίρομαι λοιπόν που ήρθα εδώ. Σε ένα θετικό κλίμα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το Made in Europe. Ε, είναι ωραίο σήμα, πρέπει να το αναπτύξουμε περισσότερο. Κάτι διαφορετικό από το Brexit. Ε, τρεις ερωτήσεις έχω. Αναφέρατε τα αυτόματα αυτοκίνητα και τα σχετικά. Πώς το βλέπετε πρακτικά να γίνεται. τα επόμενα χρόνια από πλευράς ε, όγκου επίσης. Επίσης στην ε, χώρα μου έχουμε ελλείψεις ε, στην ευρυζωνικότητα. Αλλά ακούω επίσης ότι δορυφόροι ίσως να είναι πολύ καλύτερη μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα να ακούσω την δική σας την άποψη. Έχουμε ξοδέψει πολλά λεφτά για να βάλουμε οπτικές είναι σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ αν περιμέναμε λίγο οι δορυφόροι ίσως να αποδεικνύονταν φθηνότεροι. Αυτά, επειδή μου είπατε να είμαι σύντομος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κέλλη. κύριος Σοτάξα, λοιπόν. Ε, με συγχωρείτε, έχω μια δουλίτσα εγώ αλλά ο κύριος Έλερ εδώ θα αναλάβει την ε, Προεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τις αξιόλογες παρουσιάσεις σας. Χαίρομαι για τα τόσο χαρμόσυνα μαντάτα που μας φέρατε για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα. Έχω μια τεχνική ερώτηση. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα είναι περιορισμένο Οπότε πρέπει να φροντίσουμε οι συσκευές μας ε, δεν ε, παρεμβαίνουν η μία στην άλλη, δεν δημιουργούν παρεμβολές. Γιατί αυτός ο πόρος είναι σημαντικός και κρίσιμος για, τις, για τη μελλοντική ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών. Εσείς γνωρίζετε μάλλον καλύτερα το θέμα. Έχουμε πρόβλημα με τον πόρο αυτό και η έλλειψη εξελίξεων μας εμποδίσει στην αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών. Νομίζω ότι είστε η κατάλληλη ομάδα για να απαντήσει την ερώτησή μου. Ο κύριος Τέναντ είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να μιλήσω για το Γαλιλαίο που είναι τμήμα τη Διαστημική Πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμβάλει με 1,2 δισεκατομμύρια λίρε τερλίνε στο πρόγραμμα Γαλλιαίο και στηρίξει την ανάπτυξη ικανότητων του. Και 1,2 δεν είναι ο δόλο αμεληταίο ποσό, είναι το 20% τη συνολική χρηματοδότηση του Γαλιλαίου. Και η απόρριψη των διαπραγματεύσεων τον Νοέμβριο του 2018 ε, νομίζω ότι ε, σκόπιμα οδήγησε στην ε, απέτηση για επιστροφή αυτής της ε, συνεισφοράς. Μπορείτε να μας ενημερώσετε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, αλλά λακωνικά παρακαλώ, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, όχι σε όλες φυσικά, γιατί ήταν μακροσκελής ο κατάλογος των ερωτήσεων, αλλά θα συμπληρώσουν οι συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για το διάστημα, Νομίζω ότι καταλήξαμε σε καλή διοργανική συμβαστική λύση. Αν και τελευταία στιγμή περιπλάξαν κάπως συζητήσεις, πάντως συμβαστική λύση είναι καλή. Το πρόβλημα είναι τώρα με τη χρηματοδότηση. Αν δεν έχουμε κατάλληλη χρηματοδότηση, δεν πρόκειται να λειτουργήσει το, το πρόγραμμα. Γιατί είπαμε ποια θα είναι τα ωφέλη από το διάστημα, αλλά χωρίς χρηματοδότηση δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Το θέμα του προπολογισμού είναι σημαντικό. Επίσης, διακυβέρνηση και σχέση με τον οργανισμό GSA και τον ΕΝΙΣΑ. Νομίζω ότι αυτό που προβλέπει ο νέος κανονισμός είναι μια καλή συμβαστική λύση και γίνεται μια αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των τριών οργανισμών, των τριών φορέων που είναι όλοι απαραίτητοι και θα πρέπει να, να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας αν δεν συνεργαστούμε μεταξύ μας με το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τον GSA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που δημιουργεί ο εξωτερικός ανταγωνισμός. Θέλουμε οργανωμένη και κατάλληλη σχέση μεταξύ των τριών φορέων και με τον νέο κανονισμό υπάρχει αυτή η οριοθέτηση και τώρα θα πρέπει να προσφέρουμε έργο και να την εφαρμόσουμε και εμπράκτως αυτή τη σωστή συνεργασία. Τώρα για το Κοπέρνικο. Κάποιο είπε αν έχουμε αρκετά χρήματα για το κοπένικος. Το κοπένικος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Θυμάστε ότι ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του κόσμου στην ιστορία. Και αυτή η πληροφορία στηριχθήκε σε δεδομένα που λάβαμε από το κοπένικος. Χωρίς το κοπένικος δεν θα ξέραμε και δεν μπορούσαμε να ε, συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία και όταν μιλούμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση και για την πορεία του διοξιδίου του άνθρακα, και εκεί χρειαζόμαστε το Κοπέρνικο. Έχουμε όμω αρκετό προπολογισμό στο Κοπέρνικο. Μακάρι, ελπίζουμε ότι θα έχουμε αρκετά κονδύλια. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη για το Κοπέρνικο και επανέρχομαι εδώ στη δική σα ερώτηση. Το Κοπέρνικο χρηματοδοτείται από, τη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο και από τα κράτη-μέλη του οργανισμού γιατί συμμετέχουν στη χρηματοδότηση κάποιο στοιχείο του Κοπέρνικους. Εκεί συνεργαζόμαστε και συνδυάζουμε τις προσπάθειές μας για να συγκεντρώσουμε κονδύλια για το σημαντικό πρόγραμμα που είναι το Κοπέρνικος. Ένα άλλο θέμα. Πολύ εύστοχη ερώτηση του κυρίου Σαλίνη, το θέμα του downstream. Τι θέλουμε. Θα πρέπει να εξηγήσουμε το ωφέλη του διαστήματος, αλλά και οι άλλοι τομεί να τα συνειδητοποιήσουν και αυτό δεν είναι προφανέ. Η ειδική επιτροπή είναι η κατάλληλη για να προωθήσει αυτή την επικοινωνία γιατί ασχολείστε με τη βιομηχανία, εξετάζετε τι διάφορε πτυχέ τη βιομηχανία. οπότε έχετε ρόλο να παίξετε κι εσεί. και μην ξεχνάτε και το διάστημα όταν μιλάτε για μεμονωμένους τομεί. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τι προσπάθειές μα, γιατί το διάστημα έχει κεφαλαιότητα σημασία και για την κατάντια αγορά, για την βιομηχανία, για τον ψηφιακό κόσμο αλλά έχει και κοινωνικά ωφέλη, για να μην αναφέρω τα περιβαλλοντικά που είπα πριν. Μιλήσαμε για έρευνα και διάσωση. Το γεγονό ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα πλοίο που είναι χαμένο στη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα και πολύ, με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι με το Γαλιλαίο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιο χαθεί στη θάλασσα, θα, θα βρεθεί με το Γαλιλαίο πολύ γρήγορα. Αύριο θα το βρείτε στο Twitter, θα το αποδείξουμε αύριο, θα αποδείξουμε τη χρησιμότητα του Γαλιλαίου. Βέβαια αυτό το μήνυμα δεν γίνεται αντιληπτό εύκολα και γι' αυτό και ο διαστημικός κλάδος θα πρέπει να κοιτάξει και λίγο προς τα έξω, γιατί μερικές φορές ο διαστημικός κλάδος περιορίζεται στα δικά του όρια και δεν κοιτάει λίγο έξω από, το, από τον περιορισμένο του χώρο. Επίσης, όταν μιλούμε για τη νέα διαστημική πολιτική στη ΣΥΠΑ. Ποια είναι η διαφορά. Όσοι επενδύουν στο New Space λαμβάνουν υπόψη και τι συμβαίνει σε άλλους τομείς. Δεν επικεντρώνονται μόνο στο διάστημα, αλλά συνδυάζουν και άλλους τομείς. Και αυτό ίσως θα πρέπει να το μιμηθούμε και εμείς, να το κάνουμε και στην Ευρώπη. Και μάλιστα με καλύτερο τρόπο. Και επίσης να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικούς επενδυτές στο διαστημικό κλάδο. Δεν είναι αρκετά ακόμη αυτά τα ιδιωτικά κεφάλαια. Θέλουμε φυσικά και δημόσια κονδύλια, εννοείται, αλλά και ιδιωτικά κεφάλαια, που θα είναι σημαντικό και για την ε, οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θέλουμε περισσότερε ιδιωτικέ επενδύσει και στο διάστημα. Αυτά και ο συνάδελφο θα συμπληρώσει αργότερα. Η πιο δύσκολη ερώτηση είναι το ισοδύναμο του Buy American Act, δηλαδή ένας νόμος για το αγοράστε ευρωπαϊκά. Αυτό είναι παλιό αίτημα το συζητήσαμε και για τις δημόσιες προμήθειες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφορά μόνο το διάστημα. Και είναι κάτι που όντως δεν συζητήθηκε ποτέ σοβαρά και δεν έγινε δεκτό στην Ευρώπη. Πιστεύουμε πάντως ότι όταν είμαστε, όσο πιο ανοιχτοί είμαστε, τόσο πιο ανταγωνιστικοί γινόμαστε. Θα πρέπει όμως ε, να είμαι και εγώ ανοιχτό και έντιμος και ειλικρινής απέναντί σας. Μιλάμε για το Γαλιλαίο, αλλά υπάρχει μια διάσταση, μια πτυχή ασφάλεια στο Γαλλιαίο. Οπότε μπορούμε να συνεργαστούμε μόνο με εταιρείε που έχουν την έδρα του στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ε, εμπιστευτούμε κάποιον από τρίτη χώρα και να τον εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα ε, ασφάλειας σαν του Γαλιλαίου. Μπορεί να μην έχουμε τον Buy Europe, αλλά ακριβώς επειδή το Γαλιλαίο έχει κάποιες πτυχές ασφάλειας, αναγκαστικά αγοράζουμε από εταιρείε με ευρωπαϊκή βάση. Πάντως δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο εφάμιλο με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο συνάδελφος θα απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Μία σύντομη απάντηση στην ερώτησή σας. Στην ερώτησή σας κύριε Σαλίνη για το πώς θα εξασφαλίσουμε καλύτερη μόχλευση του δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Από τη σκοπιά του οργανισμού μας, του GSA, έχουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και θεωρούμε ότι το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη δεν αρκεί από μόνο του. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δρομολογήσουμε και άλλα προγράμματα. Έχουμε ένα άλλο σχέδιο, το Κάνταλης, που ήδη φέρνει κάποιες ιδέες και προϊόντα πιο κοντά στην αγορά. Σήμερα το Horizon 2020 και στο μέλλον το Horizon Ευρώπη είναι η πρώτη γενιά. Θέλουμε και σχέδια δεύτερης γενιάς που θα φέρουν τα προϊόντα πιο κοντά στην αγορά. Αυτό είναι μία πρόταση. Άλλη είναι να προωθήσουμε επιχειρηματικά κεφάλαια στον διαστημικό τομέα. Venture capital, γιατί υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τέτοια επιχειρηματικά κεφάλαια, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Και αυτό που βλέπουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ότι θα πρέπει να βαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Και ο οργανισμό GSA έχει την τεχνογνωσία που, που χρειάζεται σε αυτόν τον τομέα που έχει ιδιαίτερα χρηματοοικονομικά, χρηματοπιστωτικά χαρακτηριστικά. Επίση, υπάρχει μια αγορά που θα πρέπει να αναπτυχθεί. Και εδώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο αγορά του κρατικού τομέα, του δημόσιου τομέα, που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και καλός πελάτης για τον GNSS. Θα πρέπει λοιπόν να προσελκύσουμε το δημόσιο τομέα και εκεί θα μπορούσαν να επικεντρωθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το έγκνος, λυπάμαι αν δεν ήμουν σαφής πριν. Όχι, ο οργανισμός GSA σίγουρα δεν παίζει κανένα ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος του έγκνος. Αυτός είναι ο ρόλος της, Ευρω... Ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο GSA ασχολείται με την παροχή επιχειρήσεων και υπηρεσιών σε ό,τι αφορά το έγνος. Και το ίδιο ισχύει και για το Γαλιλαίο. Όχι με την ανάπτυξη συστημάτων όμως. Ο κύριος Στοσενόφσκι ρώτησε τι ακολουθεί. Σε ένα μισό χρόνο από τώρα θα έχουμε πλήρη ανάπτυξη του συστήματος του, ε, του Έγνος και του Γαλιλαίου. Τώρα, τι θα γίνει στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτές, το επόμενο πι θα πρέπει να εξασφαλίζει μια συνέχεια στην παροχή των υπηρεσιών. Αυτό έχει κεφαλαιώδη σημασία. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε λοιπόν τις σημαντικές επιδόσεις του συστήματος. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και τις, την εξέλιξη στην αγορά. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα εργαλεία και άλλα επίπεδα επενδύσεων και θα πρέπει να συνδυάσουμε διάφορες τεχνολογίες. Το GNSS δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο του. Θα χρειαστεί και άλλες τεχνολογίες. Τα αυτοματοποιημένα οχήματα είναι ένα καλό παράδειγμα τα αυτοματοποιημένα οχήματα του μέλλοντό θα συγχωνεύουν διάφορες τεχνολογίες. Οπότε ένα εμπειρογνώμονα του GNSS θα πρέπει να σκέφτεται λίγο ευρύτερα και να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Ε, μιλήσατε για τα διόδια. Έχουμε περίπου 60% του GNSS στα διόδια που στηρίζονται στο GNSS δηλαδή. Και εδώ το Έγνος και το Γαλλιαίο είναι σε καλή θέση με 50-60% να χρησιμοποιούνται. 50-60% των διοδίων χρησιμοποιούν Έγνος και Γαλιλαίο, οπότε υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Μπορούμε όμως να καταργήσουμε τελείως το επίγειο σταθμό και να χρησιμοποιούμε μόνο δορυφορικά στοιχεία. Τώρα, επειδή ε, τα αυτοκίνητα έχουν μέσα δορυφορική προσέγγιση, την αυτόματη, την ηλεκτρονική κλίση το 112, έχουν ηλεκτρονικά συστήματα, οπότε χρειαζόμαστε ένα νέο κύκλωμα, ουσιαστικά ένα νέο chip, που για το GNSS θα, χρησιμο... θα εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Ένας από αυτούς θα είναι και τα διόδια. Οπότε θα αυξάνεται το κόστος ανά μονάδα του αυτοκινήτου. Αυτά και αν υπάρχει χρόνος θα απαντήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κοιτάξτε, η Επιτροπή μας ε, δεν είναι ιδιαίτερα ε, ευγενής, έχει και τη φήμη εξάλλου, αλλά δυστυχώς ε, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας ήταν ανέκαθεν υπέρ της διαστημικής πολιτικής και υπέρ της χρηματοδότησης, οπότε... Θα πρέπει τώρα να κλείσουμε με την σημερινή την συνεδρίαση, αλλά ε, στο μέλλον θα συνεχίσουμε τις επαφές μαζί σας. Σαν συνάδελφοι έχουν μείνει αναπάντητες ερωτήσεις. Ε, θα θέλαμε τις απαντήσεις σας ε, γραπτά. Γιατί τώρα έχουμε επόμενη ε, συνάντηση με το ελεκτικό συνέδριο. Οι αντιπρόεδροι έχουν χαθεί. Ε, όχι, όταν ο πρόεδρος δεν είναι εδώ, αντιπροεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Εάν οι αντιπρόεδροι δεν είναι εδώ, πρέπει να αναλάβουν οι συντονίστες. Αν οι συντονίστες δεν είναι τα μέλη και αν τα μέλη δεν είναι, τότε σβήνουμε τα φώτα και πάμε σπίτια μας. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ στο Προεδρείο. Please have a now we next topic of the agenda. We are very pleased to see the Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, με πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε το ελεγκτικό συνέδριο στο Κοινοβούλιο. Είστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι. Είναι αρμοδιότητά μας να ελέγξουμε ε, την Κομισιόν και τις δραστηριότητες της ε, σήμερα θα μας παρουσιάσετε την ειδική έκθεση για την παραγωγή ε, ηλεκτρισμού τα παλιότερα μέλη ίσως θα την ξέρετε από το όταν διατελέσει και γίνει Ευρωβουλευτής και τώρα είναι υπεύθυνη του δεύτερου τμήματος για ε, ε, ε τον έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ στην Ευρωπαϊκή, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά στην ε, Ήτρε. Δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να παρουσιάζουμε τις εκθέσεις μας, αλλά σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία ε, όσον αφορά το τοπίο της ενέργειας και του κλίματος. Θα χρησιμοποιήσω εδώ την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, για να μιλήσω για ένα project που προετοιμάζεται και που θα δημοσιευθεί σύντομα και που μπορεί δυνητικά να ενδιαφέρει την Επιτροπή σας, όπως είναι η πρωτοβουλία της Κομισιόν για ψηφιοποίηση του Ευρωπαϊκού ε, της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Industry 4.0 όπως αποκαλείται ε, σύντομα θα ε, κυκλοφορήσει και για του χρόνου θα έχουμε τις υποδομές για ηλεκτρική φόρτιση. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για την παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω της αιωλικής και της ηλιακής ενέργειας. Ε, συνήθως ε, εκείνος που έχει συντάξει την έκθεση είναι αυτός που ε, παρουσιάζει την έκθεση, όμως ο κύριος Πούφελ έχει ήδη φύγει από το ηλεκτρικό συνέδριο και γι' αυτό τον αντικαθιστώ εγώ. Δύο λόγια ε, εισαγωγικά για την αιωλική και ηλιακή ενέργεια στην Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα διότι αυξήθηκε κατά 400% και 8.000% ανάμεσα στο 2005 και το 2017 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Και μέχρι το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 8,8 δις σε project για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου ανάπτυξη και του Ταμείου Συνοχής. 922 εκατομμύρια για την αιωλική ενέργεια και 2,9 δις για την ηλιακή ενέργεια στήριξη των, ε, τα σχέδια μάλλον αυτά ε, προσέφεραν εγγύησει για τιμέ για πιστοποιητικά για την περίοδο 2021 με 27. Η Κομισιόν προτείνει γύρω στα 71,8 δις ευρώ για επιχειρήσεις που στηρίχουν, ζουν ε, στόχους για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της ε, της, του ηλεκτρισμού μάλλον ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γι' αυτό και ελέγχουμε πώς δαπανώνται αυτά τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει εθνικά στόχους, έχει θεσμοθετήσει εθνικούς στόχους για την θέρμανση και τις μεταφορές για το 2030, όμως για το 2030 καταλήφθηκαν οι εθνικοί στόχοι και τέθη ένας νέος ευρωπαϊκός στόχος. Εμείς, εν συντομία, αξιολογούμε την πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των στόχων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξετάζουμε αν η οικονομική στήριξη για την παραγωγή ηλεκτρισμού από νεολική και ηλιακή ενέργεια είναι αποτελεσματικό. Θα δώσω τώρα το λόγο, αν επιτρέπετε, το λόγο στη Χρυσούλα Λατοπούλου που είναι επικεφαλής ε, αυτής της προσπάθειας και θα σα παρουσιάσει την έκθεση. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Σίτρη, κυρίε και κύριοι, πέρυσι τον Ιούνιο δημοσιεύσαμε μια έκθεση για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αυτό του ηλεκτρισμού που προέρχεται από την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια. Η έκθεσή μας ε, συνάντησε μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ ήμουν επικεφαλής και δίπλα μου είναι ο κύριος ε, διαχειριστής ε, που επέβλεψε τους ελέγχους. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τα πορίσματα και τις συστάσεις της έκθεσής μας και στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Η νομική βάση πίσω από τον έλεγχο αυτών ήταν η οδηγία του 2008 κυρίως, που είναι γνωστή ως RED 1. Επίσης αναλύσαμε την αναθεωρημένη ε, ε, οδηγία που υιοθετήθηκε το 2018 το Δεκέμβριο και είναι μία από τις έξι ε, οδηγίες που συναποτελούν τη δέσμη για την καθαρή ενέργεια. Από το 2005 μέχρι το 2017 το μερίδιο των ανανεώσιμων στην παραγωγή ενέργειας διπλασιάστηκε από το 15% στο 31%. Αυτό οφείλεται σε μια άνευ αύξηση των όγκων ηλεκτρισμού που προέρχονται από την αιωλική ενέργεια επί 400% και από την ηλεκτρική ενέργεια κατά επί 8.000% την ίδια περίοδο, την ίδια χρονική περίοδο. Στο δεξί γράφημα, στη διαφάνεια, βλέπετε την εξέλιξη του μείγματος ε, ανανεώσιμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28 κράτη-μέλη. Ενώ αριστερά βλέπετε πως ιστορικά η ζήτηση ηλεκτρισμού παραμένει στα ίδια επίπεδα. Επίσης να τονίσουμε από το 2015 αυτές οι δύο τεχνολογίες, αιωλική και ηλιακή, από κοινού περνούν ξεπερνούν την ετήσια παραγωγή της υδροελεκτρικής ενέργειας που επισήμως παραμένει στα ίδια επίπεδα. Αυτό οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η αύξηση του ηλεκτρισμού που προέρχεται από την ολική και από την ηλιακή ενέργεια είναι καταρχάς η μείωση του κόστους της τεχνολογίας και στους δύο τομείς και δεύτερον τα κίνητρα που έδωσαν τα κράτη-μέλη που ήταν το κύριο θέμα της δικής μας έκθεσης. Η μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια ε, με μεγάλη ακρίβεια ε, φαίνεται από την εξέλιξη του δίκτυ κόστους ηλεκτρισμού. Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιείται από την βιομηχανία για να φαίνεται και να αξιολογείται το κόστος ε, παραγωγής ηλεκτρισμού από παραδοσιακές πηγές ή από τις ανανεώσιμες. Το γκρίζο, το γκρίζο ε, δείχνει το κόστος παραγωγής από ρηκτά καύσιμα και βλέπουμε ότι έχει μειωθεί η η χρήση των παραδοσιακών αυτών ε, εκπομπών. Έχουμε μείωση του κόστους των ε, ε, των ηλιακών συσσωρευτών και γι' αυτό η αιωλική και η, ηλεκτρική η ηλιακή ενέργεια έχουν καταστεί φθηνότερες πηγές παραγωγής του ηλεκτρισμού. Κοστίζει μάλιστα ο ηλεκτρισμός τους πολύ χαμηλότερα από το κόστος ε, της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ε, ορυκτά καύσιμα. Τώρα έχουμε εδώ την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνοντας το μερίδιο των ανεώσιμων πηγών ε, ε, ενέργειας. Το 2017 το 17,5% του 20% που είναι ο στόχος για το 2020 είχε επιτευχθεί. Το 2005 το σημείο κίνησης ήταν 9,1%. 11 από τα 28 κράτη-μέλη έχουν ήδη ανταποκριθεί στους εθνικούς τους στόχους, γιατί αυτοί, όπως ορίζονταν αυτοί από την οδηγία RED 1. Είναι η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Δανία, η Εστονία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Ωστόσο, οι υπόλοιποι 17 δεν είναι βέβαιο πως θα επιτύχουν να ε, ε, επιτύχουν, τους στόχους. Χαμηλό κίνδυνο αντιμετωπίζουν η Ελλάδα, η Λετωνία και η Αυστρία και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό ε, τα μέτρα που στοχεύουν τις ανανεώσιμες. Μεσαίο κίνδυνο διατρέχουν το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία εκείνοι πρέπει να αυξήσουν το μερίδιό τους στη βάση. Με ρυθμό μάλλον ε, ε, ταχύτερο. Σοβαρό κίνδυνο διατρέχουν οι κάτω χώρε, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και η Πολωνία, γιατί το μερίδιο που λείπει είναι εξαιρετικά μεγάλο για να καλυφθεί μέχρι το 2020. Αν προσθέσουμε τους 11 που ήδη έχουν πετύχει τους στόχους τους και τους 3 που διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο, συμπεραίνουμε ότι τα μισά κρατημέλη κινδυνεύουν να μην παράγουν αρκετή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους 2020. Αυτό σημαίνει πως ανησυχούμε για το κατά πόσο τα αποτελέσματα εκείνων που, έχουν, που έχουν ξεπεράσει τους στόχους θα ε, καλύψουν αυτούς που δεν τους έχουν φτάσει ώστε να φτάσουμε γενικά στο στόχο του 2020. Εμείς συστήνουμε στο να εστιαστεί η προσοχή για να, στο να κλείσουν τα χάσματα για, το 2000, για τους στόχους του 2020, να ξανασκεφτούμε το σχεδιασμό για την αιωλική και την, ηλεκτρική, και την ηλιακή ενέργεια και επίσης να να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές ε, ε, ε δικτύων. Έχουμε βέβαια συγκεκριμένες ε, αδυναμίες ε, και, αλλά και ισχυρά σημεία. Η οδηγία δίνει συγκεκριμένους στόχους αλλά και συγκεκριμένες διαδρομές για τα κράτη-μέλη. Υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ορίσουν στρατηγική από το 2010 μέχρι το 2020 όπως έπρεπε ε, να καθορίσουν πορείες και να εφαρμόσουν μέτρα για να επιτύχουν τους στόχους τους. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι οι προθεσμίες που ορίζονται από την Οδηγία ε, Στατιστικών Ενέργειας ώστε οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να δίνουν τα στοιχεία στη Eurostat είναι πολύ μακρές για να επιτρέπουν ε, την λήψη υπόψη. Δηλαδή, μόνο το 2022 θα ξέρουμε αν τα κράτη-μέλη έχουν πετύχει τους στόχους του 20. Επίσης, η οδηγία RED 1 ε, περιορίζει την εντολή της Κομισιόν στην παρακολούθηση μιας διετούς πορείας. Έτσι, η Κομισιόν δεν μπορεί να καταλάβει αν το κράτος μέλος ε, ε, ακολουθεί την πορεία που του έχει προδιαγράψει. Άρα λοιπόν το η οδηγία ΡΕΝΤ-1 έχει παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά το νομικό πλαίσιο δεν, δεν προβλέπει έγκαιρη αναφορά ή έγκαιρη ε, εντολή για την Κομισιόν ώστε να ανταποκριθεί, ε, να μπορέσει μάλλον να ε, καλύψει η Κομισιόν την αργή πρόοδο. Τα στατιστικά στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να βελτιωθούν και η χρονική του εγκυρότητα. Γι' αυτό και ο κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε από τους 11 μήνε να περάσουμε στου 9 μήνε αναφορά. Το πιο σημαντικό τμήμα της έκθεσής μας αφορά την ανάπτυξη της αιωλικής και της ηλιακής ενέργειας στα κράτη-μέλη. Για τον έλεγχο εξετάσαμε την ε, πολιτική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, στην ενέργεια, την Ελλάδα, την Ισπανία και ε, την Πολωνία. Έχουν δοθεί λοιπόν κίνητρα και από τότε το μερίδιο της αιωλικής ενέργειας στην συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού διαρκώς αυξάνεται γραμμικά με την εξαίρεση της Ισπανίας όπου η δυνατότητα, η απόδοση μάλλον έχει σταθεροποιηθεί από το 1913. Ενώ στην, ε, στην Ισπανία και στην Ελλάδα επίσης έχει σταθεροποιηθεί η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ε, λόγω μέτρων που ελήφθησαν για να καταπολεμηθεί αρχική υπερβολικά μεγάλη παραγωγή. Η Πολωνία όμως έχει μείνει στάσιμη γιατί εκείνη δεν έθεσε εφιλόδοξους στόχους για την ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο, Οι επενδύσεις στην ολική και στην ηλιακή ενέργεια ήταν υπερβολικά ε, κερδοφόρες ε, και γι' αυτό και έγιναν πολύ μεγάλες ε, επενδύσεις σε αυτήν. Είχε πολύ, είχαν πολύ ελκυστικό ποσοστό απόδοσης, πολύ υψηλότερο από τα δεκαετή κρατικά ομόλογα. Η στήριξη καλύφθηκε είτε από τους καταναλωτές όπως στη Γερμανία, είτε από τους φορολογούμενους μέσω του εθνικού ε, προϋπολογισμού στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Έτσι, ε, ψηλά επίπεδα ε, ε, στήριξης, στήριξης οδήγησαν σε ψηλότερες τιμές και στον του ηλεκτρισμού και συνέβαλαν στα εθνικά ελλείμματα. Όταν τα κράτη-μέλη να μειώνουν το επίπεδο στήριξης, η, επηρεάστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών. Επίσης θεωρήσαμε πως τα, οι ανανεώσιμες πηγές παρεμποδίζονται από ανεπαρκείς ε, πληστηριασμούς ώστε να δοθούν νέες δυνατότητες απόδοσης για τις ανανεώσιμες. Τα κράτη-μέλη επίσης ορίζουν αυστηρές προδιαγραφές, ειδικά για τη συμμετοχή των πολιτών ως καταναλωτών ή μέσω οργανώσεών τους. Τέλος, είδαμε, διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν μηχανισμούς ε, συνεργασίας, αλλά όχι ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη προθυμία. Γι' αυτό και η ενεργειακή αγορά παραμένει κατακαιρματισμένη. Συμπεράναμε ότι οι διορθωτικές ενέργειες των κρατών μελών ώστε να εξασφαλίσουν το βάρος προς τους καταναλωτές και τον εθνικό ε, προπολογισμό συνέβαλε σε, σε, σε ε, επιβράδυνση της αγοράς. Επίσης, ε, θα πρέπει να γίνουν ε, επενδύσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε τους επόμενους στόχους του 2030. Συστήνουμε στην Επιτροπή να σχεδιάσει ε, επαρκείς επιλογές, να εντοπίσει τα κατημέλη που δεν έχουν σχεδιάσει αρκετούς πληστηριασμούς και να παρακολουθεί και να αναφέρει τα αποτελέσματα των πληστηριασμών αυτών. Τέταρτο πόρισμα αφορά άλλα προσκόμματα που καθυστερούν την πλήρη εφαρμογή των, της και, και ηλιακής ενέργειας. Ε, περιορισμούς στις χωροταξικούς κανόνες και χρονοβόρες διαδικασίες. Ιδιαίτερα με τους περιορισμούς χωροταξικούς εννοούμε ότι βρήκαμε περιφέρειες που έχουμε ελάχιστη επιτρεπόμενη ε, απόσταση ε, που είναι, για τις ανεμογεννήτρες είναι 10 φορές το συνολικό μήκος της ανεμογεννήτρες, δηλαδή μπορεί να φτάσει και 2 χιλιόμετρα. Στη Γερμανία ο αντίκτυπος του μέτρου ήταν να μειώσει το, τη γη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αιωλικά πάρκα ε, περίπου 0,3% σε σχέση με την προβλεπόμενη περιοχή γύρω στο 3%. Με το μέτρο αυτό στην Πολωνία η επιλέξιμη γη για τις επενδύσεις μειώθηκε στο 0,1% της εθνικής επικράτειας σε σχέση με το 2,6% που ήταν αναμενόμενο. Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες, τα κράτη-μέλη όρισαν ανώτατα χρονικά όρια για τη συγκέντρωση όλων των αδειών ε, για να κατασκευαστεί ένα αιωλικό πάρκο ή πάρκο αιωλική και φωτοβολταϊκή ενέργειας, κάτι που δεν έγινε όμω στην Ισπανία και την Ελλάδα. Ε, στις δύο αυτές χώρες μπορεί να χρειαστεί και μία εφταετία για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο. Ενώ κανονικά πέντε χρόνια θα ήταν αρκετά για την εφαρμογή του. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ε, περιοριστικοί κανόνες χωροταξίας περιορίζουν την ε, ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων και χρονοβόρες γραφειοκρατικέ διαδικασίες περιπλέκουν το ρυθμιστικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για την αιωλική ενέργεια. Συστήνουμε λοιπόν απλούστευση των διαδικασιών και δημιουργία πιο πρόσφορου ε, περιβάλλοντος για την ενθάρρυνση των επενδύσεων πέμπτο πόρισμα για το δίκτυο. Οι επενδύσει στο δίκτυο καθυστέρησαν αισθητά και στι τέσσερι στις τέσσερις χώρες που ε, επισκεφτήκαμε, ειδικά στη Γερμανία. Λιγότερο το 10% της ε, σχεδιαζόμενης επέκτασης του ε, σχεδίου είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 2017. Βέβαια, Εξαιτία αυτή τη λοιπού ανάπτυξη έχουμε χαμηλέ ροέ ενέργεια με τι γειτονικέ χώρε, ενώ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πλεόνασμα στι μεταφορέ. Επίση, έχουμε κάποιε ανεπάρκειε του δικτύου που εμποδίζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε, χώρες, σε περιοχές που έχουν μεγάλο δυναμικό αιωλικής ενέργειας, στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, γιατί δεν μπορούν να εγκαταστήσουν νέα σχέδια ΑΠΕ. Επίσης, για να υλοποιηθούν ε, οι στόχοι του 32% για το 2030 χρειάζεται 55% μερίδιο της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ. Σήμερα ο τομέας ενέργειας ε, συμβάλλει κατά 31% στους στόχους του 2020, κάτι που ήδη δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα για το δίκτυο. Και για να πάμε από το 31% στο 55% που απαιτείται, ε, προϋποθέτει κατεπηγόντως επενδύσεις. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι καθυστερήσεις στις επενδύσεις του δικτύου και στις διασυνδέσεις υποδομής εμποδίζουν την ανάπτυξη ΑΠΕ και την ε, δημιουργία συνεργειών μεταξύ των κρατών μελών και προτείνουμε προώθηση επενδύσεων στις υποδομές δικτύου και στις γραμμές διασύνδεσης. Μόνο έτσι θα διορθωθούν οι ανεπάρκειες και θα εξασφαλιστεί κατάλληλη υποστήριξη του Ταμείου Συνοχής και του Περιφερειακού Ταμείου για να αντιμετωπιστούν οι κλιματικέ αλλαγέ χάρη στην ανάπτυξη δικτύου, στη σωστή διαχείριση και στη δημιουργία γραμμών διασύνδεση. Έκτο συμπέρασμα, έκτο πόρισμα, την, αφορά την οδηγία αναδιατύπωση και τον κανονισμό διακυβέρνηση του πακέτου καθαρή ενέργεια. Σε σχέση με την πρώτη οδηγία για, τους, για τις ΑΠΕ, το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο στηρίζει περαιτέρω την εξάπλωση των ΑΠΕ. Απαιτεί κάποιες βελτιώσεις στο σχεδιασμό και τη σταθερότητα των σχεδίων στήριξη, προωθεί την αυτοκατανάλωση τη ενεργειακή κοινότητες, απαιτεί τη δημιουργία μόνο απευθυντική θηρίδας για το συντονισμό τη αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και θα την θέσπιση χρηματοδοτικών μέσων και επίσης ο κανονισμός διακυβέρνησης ε, επεκτείνει την ε, εντολή παρακολούθησης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμη κάποιες αδυναμίες. Ε, το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι η εθνική στόχη της πρώτης οδηγίας ΑΠΕ ήταν πιο σημαντικός, ε, το πιο σημαντικό έναυσμα για τις ε, πολιτικές ΑΠΕ και τις επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Η δεύτερη οδηγία ΑΠΕ αντικαθιστά τους εθνικά δεσμευτικούς στόχους με ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς στόχους τουλάχιστον 32%. Αυτό ενέχει το κίνδυνο είτε τα κράτη-μέλη να είναι καλοί μαθητές σε ό,τι φορά τους ΑΠΕ, αλλά και άλλα κράτη να μείνουν πίσω. Οπότε θα υπάρξει μεγάλο χάσμα σε ό,τι φορά τη χρήση των ΑΠΕ. Επίσης, ε, δεν γίνεται έγκυρη ενημέρωση, υποβολή εκθέσεων. Δεν έχει διορθωθεί ακόμη αυτό. Και να μην ξεχνούμε ότι η δεύτερη οδηγία ΑΠΕ θα πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Και τα τέσσερα μέλη, κράτη-μέλη που εξετάσαμε μετέφεραν με καθυστερήσει την πρώτη οδηγία ΑΠΕ. Και η Πολωνία καθυστέρησε έως και τέσσερα έτη για τη μεταφορά στην Εθνική Ενωμή Οπότε αναγνωρίζουμε ότι η οδηγία ΑΠΕ και ο κανονισμός της διακυβέρνησης έχουν μέτρα που συμβάλλουν σε καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον. Βέβαια, η έλλειψη εθνικών στόχων σε συνδυασμό με την αδυναμία να αντιμετωπιστούν τα προηγούμενα μειονεκτήματα σε σχέση με την μία εγκαιρή ενημέρωση ε, θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των νέων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030. Θα πρέπει να βελτιωθεί ο έλεγχος ώστε να αντισταθμιστεί η έλλειψη εθνικών δεσμευτικών στόχων και να μεταφερθεί η οδηγία στην Εθνική Τάξη εγκαίρως, ε, σωστά και εμπρόθεσμα. Και φτάνω στο τέλος της παρουσίαση της ειδική έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ε, ευχαριστώ για την προσοχή και περιμένω τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα εδώ πέρα την αίθουσα, δεν υπάρχει συντονίστρια. Έχω μια σύντομη ερώτηση για τη μεθοδολογία για το έβρεμα υπαριθμών 4. Αναφερθήκατε στην απόσταση οικισμών που μειώνει έτσι τις περιοχές οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν απ' έξω όσον γνωρίζω στην Ευρώπη και στην Πολωνία η απόσταση που απαιτείται από το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα εθνικά παρκά είναι ακόμη μεγαλύτερη ε, από τους οικισμούς. Αυτό λίγο δεν ε, άλλαξε τα ευρήματά σας γιατί εξορισμού η απόσταση των εγκαταστάσεων αυτών Ε, δεν είναι πάνω από 50% από τους ανθρώπινους οικισμούς. Ε, καθορίζεται, παραδείγματος χάρη, από την απόσταση από πουλιά που αναπαράγονται, που είναι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται, δηλαδή, είναι, μεθοδολογία, είναι αποτυχία της μεθοδολογίας, γιατί συνεπίες έχει. Ή απλώς κάνω λάθος. Παρακαλώ. Κυρία Κουταγιάρ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την μελέτη σας και για το ότι ήρθατε εδώ. Θα ήθελα να εστιάσω σε μία από τις συστάσεις που κάνετε λέτε την ανάγκη να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες για την παραγωγή από ΑΠΕ και λέτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος από την επαφή με την δημόσια διοίκηση. Το πρώτο φορά στον κίνδυνο του να δραστηριοποιούνται σε μια χώρα όπου το συγκεκριμένο έργο γίνεται και το δεύτερο είναι ο κίνδυνος ε, του να επενδύσουν ε, και η γραφειοκρατία μία συγκεκριμένη χώρα. Η αρχική φάση ενός ε, έργου μπορεί να αποτελεί ως και 10% του έργου, δηλαδή να δουν την πολυπλοκότητα της εθνικής διοίκησης, να βρουν το κατάλληλο μέρος, να πάρουν τις άδειες κτλ. Εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ε, οι χώρες θα καταφέρουν να επιτύχουν τους ε, στόχους, ειδικά εν ώψη των στόχων του 2030, θεωρώ ότι θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε την ε, φάση ανάπτυξης ενός έργου και να επενδύσουμε περισσότερο. Και κάποιοι έχουν δει την πιθανότητα να τα κάνει αυτά η δημόσια διοίκηση, δηλαδή να υπάρχει μια φάση δημοσίων προμηθειών στην πρώτη φάση και έτσι θα μειωθούν οι κίνδυνοι και θα αυξηθούν οι επενδύσεις και θα αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δημιουργώντας θέσεις εργασίας αλλά και θα διαβεβαιωθούν οι πολίτες για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο τέτοιων έργων. Εσείς ε, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει περισσότερες ΣΔΙΤ για να εγγυηθεί αυτή την διαδικασία και ότι μια δημόσια διοίκηση θα πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνη για την αρχική φάση ενός έργου και αν ναι, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να επιταχύνει αυτές τις διαδικασίες για να επιτύχει τους στόχους της η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να βοηθήσουμε αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ για το ερωτηματικό σας. κύριος Ρόμπ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές ε, τις ομιλήτριες ε, για την παρουσίαση της μελέτης βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών, άλλες παράγουν περισσότερη ενέργεια, άλλες λιγότερη. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η ΑΠΕ είναι ενέργεια του μέλλοντος, η οποία παράγεται δωρεάν. Πρέπει απλά να δούμε τις δομές και τις υποδομές για να παράγεται με σωστό τρόπο. Βλέπετε επίσης ότι η τεχνολογία θα μας επιτρέψει να παράγουμε ηλεκτρισμό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Γιατί κάποιες χώρες παράγουν 20% και παραπάνω ενώ άλλες ε, έχουν ε, ε, πολύ χαμηλότερο 1%. Μετά, μία άλλη ερώτηση. Θεωρώ ότι το κοινό επιζητά περισσότερα τέτοια έργα, αλλά βλέπουμε ότι κάποιες χώρες, όπως η δική μου, ας πούμε, η Λιθουανία, ε, τα πήγαινε καλά σύμφωνα με τη μελέτη σας, αλλά βλέπουμε επίσης ότι και το κοινό δεν κάνει πολλά για ε, να παράγει περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια. Όμως η χώρα μου δεν αγοράζει τον ηλεκτρισμό. Δηλαδή τι γίνεται. Ε, υπάρχει κάποιος παραγωγός που χρησιμοποιεί την ενέργεια, αλλά πρέπει να την δωρήσει στο δίκτυο. πώς αυτό είναι εμπόδιο στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και τι λύση θα μπορούσε να βρεθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχω 6-7 άτομα εδώ στον κατάλογο. Πρέπει να τελειώσουμε 5 παρα 10 και για να έχουμε κάποια απάντηση θα ήθελα να περιορίσω τις ερωτήσεις στο ένα λεπτό. Και μετά από αυτό, εντάξει θα έχετε όλη την ε, ευκαιρία σας, ε, αλλά πρέπει να απαντήσουν και οι κυρίες. Ε. Λοιπόν, ο κύριος Γκρούτλερ κατόπιν. Sorry, my name is Grudler. Grudler ονομάζομαι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά. Σύντομα, ερώτηση. Η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια είναι απαραίτητε ε, και μας παρουσιάζεται τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Συγκεκριμένη ερώτηση. Αν η αιχμή της παραγωγής σπάνια ανταποκρίνεται ε, στην αιχμή κατανάλωσης στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ΑΠΕ ε, δεν μπορούν ε, να αποθηκευθούν. Οπότε στη μελέτη σας εξετάσατε πώς οι χώρες συμπληρώνουν την έλλειψη ΑΠΕ κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες της μέρες και από τι το αντικαθιστούν από την ε, από συνδυασμένο κύκλο από ορυκτά καύσιμα και υπάρχει δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιμείνουμε στην χρήση υδρογόνου χωρίς ε, άνθρακα, ώστε να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια και να μπορούμε να παράγουμε ενέργεια ε, ηλεκτρική τις ε, ώρες εκείνες που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος blackout, κατάρρευσης του δικτύου. Ευχαριστώ. Κύριος Φουλσάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Νομίζω η τελευταία σύσταση ότι πρέπει δηλαδή να μεταφραστεί ο γενικό στόχο του 32% σε συγκεκριμένου στόχου ανά χώρα είναι προφανής αλλά πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να γίνει αυτό για τους στόχου του 2030 το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να επεκταθείτε στην σύσταση για τα στατιστικά στοιχεία. Αν προξενεί εντύπωση το ότι έχουν καθυστερήσει δύο χρόνια από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Οπότε, τι άποψη έχετε για τα στατιστικά στοιχεία. Μπορούμε να έχουμε στατιστικά στοιχεία σε ε, ε, επίκαιρα στατιστικά στοιχεία ανα πάσα στιγμή ή τι άλλο μπορεί να γίνει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Φλέγκο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό να επισημάνουμε είναι φυσικά όλοι είμαστε υπέρμαχοι των ΑΠΕ, όλοι είμαστε υπέρ της ολικής ενέργειας, υπέρ της ηλιακής ενέργειας, αλλά το θεμελιώδες ερώτημα που ανακύπτει είναι η ανταγωνιστικότητα. Οπότε ρωτώ, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ενισχύσουν την ε, ανταγωνιστικότητα της οικονομίας τους ε, με λήψη υπόψη της οικολογίας, ε, αλλά να μην χάσουμε λόγω της οικολογίας την ανταγωνιστικότητά μας και να μην θυσιάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας ε, στις ΑΠΕ και να μην επωφεληθούν από αυτή την αντική μας απόλυτη ανταγωνιστικότητα η Κίνα, η Ρωσία ή άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πάουλους, ε, σας ευχαριστώ. Υποθέτω ότι θα μας στείλετε τις διαφάνειες. Ωραία, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, η απόσταση από τα πτηνά που ζευγαρώνουν δεν είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ίσχυε αυτό, αν υπήρχαν ξεκάθαρα κριτήρια, δεν θα αποφάσιζαν ε, κατά περίπτωση σε κάθε έργο και καλό θα ήταν να υπάρχουν τέτοια κριτήρια. Έχω μία ερώτηση για την ε, διαφάνεια για τα ορυκτά καύσιμα. Υπάρχει εκεί ένα φάσμα που δώσατε ένα ευρώ. Έχουν εντύπωση πως ε, και τα νέα και τα υφιστάμενα ε, περιέχονται εκεί. Για ποια τιμή ανανεώσιμων είναι αυτό η σημερινή τιμή ή η τιμή του 2015 γιατί όπως αναφέρθηκε έχει πέσει πολύ επίσης. Θεωρείτε ότι οι πληστηριασμοί είναι πιο αποτελεσματική για να επιτύχουμε εγκαίρως τους στόχους μας σε σχέση με τις εγγυημένε τιμές και αν ναι γιατί, ε, με την ε, Γερμανία από όταν πέρασαν στους πληστηριασμούς έχουν μειωθεί πάρα πολύ η πάροχη, η ποικιλομορφία τους δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Κύριος Γκονζάλες. Ευχαριστώ ευχαριστώ και το Ελεκτικό Συνέδριο για την εξαιρετική έκθεση που κάνει μια πολύ άρτια διάγνωση της κατάστασης. Συγκεκριμένες ερώτησεις. Είπατε ότι με την νέα οδηγία ΑΠΕ δεν έχουμε πια εθνικά δεσμευτικούς στόχους και θα είναι δύσκολο με ευρωπαϊκά δεσμευτικούς στόχους να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2030. Θεωρείτε ότι ο ρόλος του κανονισμού για τη διακυβέρνηση ε, μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη εθνικών δεσμευτικών στόχων. Και αν όχι, τι προτείνετε, τι συστήνετε για να ενισχύσουμε τη συμμόρφωση πέραν της σωστής εφαρμογής ε, της οδηγίας στο ε, εθνικό δίκαιο. Είπα ότι θα πρέπει να παραμείνουν τα συστήματα στηρίξης των ΑΠΕ. Είπατε όμως ότι η αιωλική και φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι όριμες οικονομικά τεχνολογίες και οικονομικά ανταγωνιστικές. Οπότε τι είδου ε, συστήματα υποστήριξης προτείνεται για αυτή την κατάσταση. Θεωρείτε ότι αυτά τα συστήματα θα πρέπει να λάβουν υπόψη και άλλες ΑΠΕ και λιγότερο όριμες τεχνολογίες ή έχετε υπόψη και άλλα προσκόμματα πέραν των οικονομικών και γραφειοκρατικών και εκεί ε, επικεντρώνεται τα στήματα στήριξης. Επίσης, ε, οι Power Purchase Agreements, τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν σε όλα αυτά. Ο κύριο Πεκάρινεν. Ε, η, παραγωγή ολικής ενέργειας είναι πολύ μετάβλητη. Και να κάνω μια σύντομη ερώτηση. Έχετε κάνει μια επισκόπηση για να εξισορροπηθεί ε, η προσφορά και η ζήτηση αυτής της παραγωγής ενέργειας με ολική ενέργεια. Τι εργαλεία υπάρχουν, τι μηχανισμοί υπάρχουν ε, σε διάφορα κράτη-μέλη για να αντισταθμιστεί αυτή η διαφορά προσφοράς και ζήτησης με τη χρήση ολικής ενέργειας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπλος. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεσή σας. και πραγματικά επισημαίνει πολλά ενδιαφέροντα που θα πρέπει να απασχολήσουν και την Επιτροπή μας. Θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις για, τις, ε, για τον ανεπαρκή αριθμό δημοπρασιών που επισημάνατε. Ποιο είναι αυτό το κόστος ε, ανεπαρκούς ε, πληστηριασμού. Ε, είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρονται η Γερμανία και η Πολωνία για χωροταξικούς περιορισμούς που δημιουργούν προσκόμματα. Κι όμως η Πολωνία έχει τεράστιες ευκαιρίες ε, με την αιωλική ενέργεια, για παράδειγμα. Μπορείτε όμως να μας βάλετε να, να ποσοτικοποιήσετε αυτή την ε, ικανότητα της Πολωνίας και τι κέρδος μπορεί να έχει από τη χρήση αιωλικής ενέργειας. Ευχαριστώ κυρία Μίλλερ. Μάλλον Μελάχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις εκπροσώπους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα σταθώ σε μια παρατήρησή σας για τους περιορισμούς στην ανάπτυξη επενδύσεων ε, στην νεολική και φωτοβολταϊκή ενέργεια. Μιλήσατε για κάποιους χωροταξικούς περιορισμούς. Για την νεολική ενέργεια σταθήκατε σε δύο χώρες και στους περιορισμούς τους στη χωροταξία. Και στις δύο περιπτώσεις ε, έχουμε την εντύπωση ότι ε, αρχικά είχαμε μια εκθετική αύξηση της αιωλικής ενέργειας και μετά μια στασιμότητα. Αλλά ε, δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε στην εθνική κυριαρχία ε, για θέματα χωροταξίας. Μπορείτε να μας καθησυχάσετε σε αυτό ότι δεν θα υπάρξει τέτοια επέμβαση. Επίσης, έχουμε μια επιβράδυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Ενώ αντίθετα έχουμε επέλαση των αλλοδαπών τεχνολογιών, κυρίως κινέζικης τεχνολογίας στις ΑΠΕ. Ευχαριστώ και περιμένω τις διευκρινήσεις σας. Και τέλος, ο κύριος Ρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε το ότι οι ανεμογεννήτριες ε, είναι πιο καθαρές για το περιβάλλον και για την υγεία αλλά γνωρίζετε τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τις επιπτώσεις ε, το, που έχουν στην υγεία και των ανθρώπων ε, και των ζώων επίσης και βεβαίως ε, ε, καταλαμβάνουν και χώρο πολύτιμο και καταστρέφουν το τοπίο. Ένα άλλο ερώτημα αναφερθήκατε στην σταθερότητα του δικτύου μας. Τον Ιούνιο στην Γερμανία είχαμε τρία ε, παραλίγο blackout ε, λόγω ε, των πάρα πολλών ανεμογεννητριών που έχουν εγκατασταθεί και βέβαια εξαρτώμεθα από την φύση. Το ερώτημά μου είναι τα λαμβάνετε αυτό υπόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, οπότε εδώ πέρα τελειώνει ο κατάλογος των ομιλητών. Μία προσθήκη, γιατί όπως σας το είπε η κυρία Πάολο, αναφέρθηκα στην οδηγία για τα οικοσυστήματα χλωρίδας και πανίδας, το FFA. Ε, λυπάμαι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. 22 ερωτήσεις ε, διατυπώθηκαν και ουσιαστικά έχουμε 7 λεπτά για τις απαντήσεις. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε τουλάχιστον ένα τέταρτο στις καλεσμένες μας, γιατί έχουμε και άλλο θέμα στην ημέρη σε διάταξη μετά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και μοιράστε τον μεταξύ σας το χρόνο. Εγώ θα κάνω μια γενική παρατήρηση για, τα, για τις ΔΙΤ και μετά με τα πιο τεχνικά θέματα θα τα παραπέμψω στους συναδέλφους. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί η μελέτη αντικτύπου της δεύτερης οδηγίας για τις ΑΠΕ κατέληξε στο στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 250 δισεκατομμύρια επενδύσεις για, τις αρχικές, για τους αρχικούς στόχους του 2030. Και σήμερα έχουμε πολύ χαμηλότερα ποσά. Οπότε αναμένουμε να έχουμε 71,8 δις για να, για να υλοποιήσουμε τους στόχους α, α, τους περιβαλλοντικούς από το ΦΕΝΤΕΡ και το Ταμείο Συνοχής. Έχουμε τεράστιο κενό λοιπόν επενδυτικό. Χρειάζομαστε και ιδιωτικέ επενδύσει για να το καλύψουμε. Ποιο ήταν ο ρόλο των ΣΔΙΤ. Είχαμε μια άλλη ειδική έκθεση, δεν ξέρω αν σα την παρουσιάσαμε, για τη συμπράξη ιδιωτικού και δημοσιοτομέα. Πάντω θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη ΣΔΙΤ, γιατί κάποια συμπεράσματα τη προηγούμενη έκθεση του Ενεκτικού Συνεδρίου προέβλεπαν ότι ε, ο συντελεστή κόστο οφέλους και η διαφάνεια ε, έχαναν κάπου. Και παρόλο που υπάρχει κάποια αξία, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ιδιαίτερα όταν μιλούμε για τέτοια αστρονομικά ποσά επενδύσεων. Μιλάμε πάνω από δια... για επενδύσεις άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα θα παραπέμψω το λόγο στους συναδέλφους, γιατί άκουσα ότι θέσατε πάνω από 20 ερωτήσεις. Ναι, θα ήταν εύκολο να τις καλύψουμε, γιατί Φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και προκαλεί ζωηρή συζήτηση. Είναι αδύνατο να κάνουμε έλεγχο στα πάντα, σε όλα αυτά που αναφέρατε. Ξεκινώ λοιπόν από αυτά που είναι εκτός της εμβέλειας του ελέγχου μας. Εμείς δεν εξετάσαμε ούτε το θέμα της κινέζικης τεχνολογίας, ούτε το θέμα των ευρωπαϊκών επενδύσεων και της μείωσής τους. Αυτό εκφεύγει το δικό μας ε, ελέγχο. Σε ό,τι αφορά τις ανεμογεννήτριες ε, και τις ε, επιπτώσεις στην υγεία ή τη θνησιμότητα των πτηνών, και αυτό είναι εκτός της έκθεσής μας. Από ό,τι πάντως διαπιστώσαμε την τελευταία διετία που ασχολούμαστε με τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία λόγω των ανεμογεννητριών. Και είχαμε και ένα πάνελ εμπειρογνωμών που μα διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν αρνητικέ επιπτώσει υγεία από τι ανεμογεννήτριε. Η θνησιμότητα των πτηνών είναι κάποιο θέμα, αλλά αν κάνουμε μια σωστή ανάλυση πού θα τοποθετήσουμε το υλικό πάρκο με τις ανεμογεννήτριες, τότε μπορούμε να παρακάμψουμε το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα του δικτύου ε, μετά από τις, ε, λόγω των ε, ανεμογεννητριών που λειτουργούν. Όντως, είναι διαλείπονο χαρακτήρα στον ΑΠΕ. Δεν υπάρχει μία αμύωτη ροή. Και αυτό όμως ε, δεν εμπίπτει στον ελεγχό μας. Πάντως αυτό που μάθαμε είναι ότι όταν έχουμε πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούμε να το πουλήσουμε στους γείτονε. Άρα απαιτούνται περισσότερες γραμμές διασύνδεσης. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη καλές γραμμές διασύνδεσης. Και ικανότητες διασύνδεσης με τις γείτονες. Οπότε μια λίστα ήταν αυτή για να παρακαμφθεί αυτή η διαλείπουσα ροή της ΑΠΕ. Σε ό,τι αφορά την ανεπάρκεια των πληστηριασμών. Με τους πληστηριασμούς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2016 δεν μπορεί να κατανεμηθεί νέα ικανότητα με τις παλιές ταρίφες. Και αυτό είναι κάτι που προκύπτει από την ανάλυση μας, γιατί η αγορά αιωλικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας είναι πια έτοιμη να μπει στην ελεύθερη αγορά, δεν χρειάζεται επιδοτήσεις. Οπότε το θέμα των, της ανεπάρκειας πληστηριασμών οφείλεται στον προγραμματισμό των κρατών μελών. Αν μια χώρα δεν θέλει να προγραμματίσει τακτικ, τακτικές δημοπρασίες ή δεν θέλει να αναπτύξει την πράσινη ενέργεια μέσω αιωλικής και ηλιακής ενέργειας. Αυτό είναι εθνική απόφαση, κυρίαρχη. Και εδώ ίσως ερχόμαστε στο πιο ενδιαφέρον Το ενεργειακό μείγμα μιας χώρας με βάση τις συνθήκες είναι εθνικό ζήτημα. Οπότε κάθε κρατος μέλος μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να χρησιμοποιήσει το μείγμα του το ενεργειακό περισσότερες ΑΠΕ ή περισσότερα ορυκτά καύσιμα. Αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ενεργειακό μείγμα και τη σύνθεσή του. Τώρα για την αποθήκευση και την παραγωγή που δεν ακολουθεί την κατανάλωση. Ούτε και αυτό εμπίπτει στον έλεγχο. Αν και πρόσφατα είχαμε πριν από δύο μήνες εκδώσει ειδική έκθεση για την αποθήκευση. Δεν θυμάμαι τον κωδικό, αλλά τον, το καλοκαίρι του 2018 τον είχαμε εκδώσει, οπότε σας παραπέμπω εκεί, στην ειδική μας έκθεση για την αποθήκευση της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία και τα, τις ειδικές στατιστικές πληροφορίες αναχώρα, η οδηγία εγκρίθηκε πολύ πρόσφατα, το Δεκέμβριο του 2018 και η απόφαση που ελήφθη είναι να μην υπάρχουν εθνικά δεσμευτικοί στόχοι. Τώρα, για τα επίκαιρα στατιστικά στοιχεία. Και εμάς μας ε, εξέπληξε γιατί η οδηγία για την ενέργεια προβλέπει 11 μήνες. Γιατί μέσα στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς τη στιγμή που μιλάμε τι, πόση ηλιακή και αιωλική ενέργεια παράγεται. Αυτά όμως τα στατιστικά στοιχεία για την ενέργεια περιλαμβάνει και άλλα θέματα, όπως τη βιομάζα ή πόσο ξύλο κάει και το χειμώνα, πόσα ξύλα χρησιμοποιήθηκαν. Και τα στατιστικά γραφεία για να συγκεντρώσουν τα στοιχεία αυτά πρέπει να κάνουν έρευνες. Και οι έρευνες είναι χρονοβόρα διαδικασία. Και οι δημοσκοπήσεις. Οπότε ζητήσαμε από τη Eurostat, συστήσαμε στη Eurostat, Eurostat να ζητήσει από τα κρατημέλη το ενδεκάμινο να το κάνουν εννιάμινο, ότι αμέσως την επόμενη χρονιά, δηλαδή στα τέλη του 2020-2021, να έχουμε τα στοιχεία για το 2020 ώστε να μην περνάει ένας χρόνος από τη λήψη των στοιχείων και την πραγματικότητα που αντικατοπτρίζουν. Τώρα, για τους Κινέζους και την ανταγωνιστικότητα και αν τα κράτη-μέλη ε, επενδύουν στην ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετική θέση σε ό,τι αφορά το δυναμικό αιωλικής και ηλιακής ενέργειας. Κάποια στιγμή όμως μπήκε και η Κίνα δυναμικά στην αγορά. Αλλά μην ξεχνάτε τι πληθυσμό έχει η Κίνα και τι πληθυσμό έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην περιμένετε το ίδιο δυναμικό με την Κίνα και δεν χρειαζόμαστε και τόσο δυναμικό. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Ε, μιλήσατε για τη διαφάνεια που αναφέρει το κόστος και το φάσμα. Δεν είναι δική μας αυτή η γραφική παράσταση. Τη δανειστήκαμε από την Ιρένα, τον οργανισμό που κάνει μελέτες για τα θέματα αυτά. 60 μέλη έχει, 27 χώρες μέλη συμμετέχουν εκεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένας από τους συμβούλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ρένα για θέματα ενέργειας. Δεν ξέρω πώς συγκέντρωσα τα στοιχεία και κατέληξα σε αυτή τη γραφική παράσταση, αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για κόστος. Και δεν νομίζω ότι ε, οι επιχειρήσει παραγωγή ηλεκτρισμού θα έρθουν τόσο εύκολα και ο θελός θα μα ε, δηλώσουν το κόστο του και τι ταπάνε του. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα απλά να συμπληρώσω κάποιε απαντήσει ε, για το πεδίο εφαρμογή. Λέμε στην έκθεσή μα ε, στην παράγραφο 16 ότι εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των 100 μελών στην επίτευξη των στόχων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Δεν έχουμε εξετάσει όλα τα θέματα που μας ρωτήσατε. Έχει λίγο επιβραδυνθεί η πρόοδος γι' αυτό και ε, κάποιες από τις ερωτήσεις που μας θέσατε ήταν εκτός ε, του δικού μας πεδίου και όσον αφορά το κόστος δεν το εξετάσαμε αυτό γιατί εστιάσαμε στην παραγωγή για τους εθνικούς στόχους από ό,τι κατάλαβα αυτό αφορούσε τη νέα RED 2. Εκεί η σύστασή μας είχε στόχο τους ισχύοντες κανόνες, δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τους νομοθέτες. Εμείς λέμε ότι μέσα στο πλαίσιο αυτών των κανόνων που ισχύουν θα έπρεπε να παρακολουθούμε καλύτερα ώστε να μπορούμε να δείξουμε εάν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο γιατί διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους στο τέλος της ε, περίοδου. Τώρα, για τη χωροταξία, αυτό που εξετάζουμε ήταν μόνο η χωροταξία αποκλειστικά και θέλαμε να δείξουμε πως οι αποφάσεις εκεί έχουν περιορίσει το χώρο που θα είναι διαθέσιμος για την παραγωγή ηλιακής ή αιωλικής ενέργειας πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο στόχος ε, αυτού του γραφήματος, ότι δεν μπορούμε από τη μια πλευρά να λέμε ότι θέλουμε να παράγουμε πολύ περισσότερο, ενώ από την άλλη μεριά μειώνουμε τις δυνατότητες ε, ε, όπου μπορούν να κατασκευαστούν δηλαδή αιωλικές, αιωλικά πάρκα ε, ή πάρκα συσσωρευτών. Πρέπει να γίνονται συνδυασμένα οι προσπάθειες. για την έναρξη δημοσίων προγραμμάτων. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε ε, για το πώς ε, οι διαχειριστικές αρχές αποφασίζουν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν τη τεχνική αρρωγή που έχουν στη διάθεσή τους για να βοηθήσουν τους ε, Ε, φορείς πόσο θέλουν να έχουν επαφές με τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα για να, όταν έχουν ιδέες ας πούμε για το ε, προσιτές ε, για να περάσουν από τα διάφορα βήματα να έρθουν σε επαφή με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Βασικά είναι εθνική απόφαση αυτό. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, η Red 2 επιχρεώνει τα κρατη να φτιάχνουν μία μόνο θηρίδα για όλα. Από το 2021 οφείλουν να φτιάξουν ένα γραφείο το οποίο αναλαμβάνει την προετοιμασία ολόκληρης της ε, ε, τεκμηρίωσης, αυτό που γίνεται ήδη στη Γερμανία. Στις 6, στους 6 μήνες στη Γερμανία μπορείς να, βρεις, να βγάλεις την άδεια, ενώ στα άλλα κράτη-μέλη ε, χρειάζεται πάνω από χρόνο. Ελπίζουμε λοιπόν πως όλα αυτά θα λειτουργήσουν. Κυρίε και κύριοι, λοιπόν, ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο και χαιρετίζω την πειθαρχία σας, ε, γιατί ε, είστε ένα σημαντικό ε, ε, σημαντική πηγή πληροφοριών για μας εδώ στο Κοινοβούλιο και τέτοιου είδους εκθέσεις πάντοτε μας είναι χρήσιμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντοτε ξέρετε έχουμε περιορισμένο χρόνο. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχετε εσείς περισσότερο χρόνο και ευχαριστώ τους συναδέλφους που περιορίστηκαν στο ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ και πρέπει τώρα να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα. Να σας ε, ευχαριστήσω λοιπόν κυρία Ιβάνοβα, κυρία Λατοπούλου και κύριο Μπρόκοπα. Θα τα πούμε πάλι σύντομα. the chair gets a little bit nervous because I'm meant to be here till quarter past. Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι θα ήμουν εδώ πέρα μέχρι τις ε, 5 παρατέταρτο, αλλά περνάμε στο επόμενο θέμα. Παρουσίαση της έκθεσης για το πρόγραμμα κλεισίματο πυρηνικών σταθμών σε Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία. Να υπενθυμίσω στου βουλευτέ πως όταν εντάχθηκαν αυτές οι χώρες δεσμεύτηκαν να κλείσουν 8 πυρηνικά εργοστάσια πριν από το τέλος της προγραμματισμένης ζωής τους. Έχουμε λοιπόν ε, τα διαφορά εργοστάσια εδώ. Να ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Γκαρίμπα, τον υποδιευθυντή της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, να μας παρουσιάσει την έκθεση που αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών για το 2018. Έχουμε 45 λεπτά. Ε, έχει έρθει. Αναμένουμε με αγωνία λοιπόν. Α, θα μιλήσετε από εκεί που κάθεστε, μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα προσπαθήσω πράγματι να σας δώσω μια εικόνα του προγράμματος. Όπως θα θυμάται θα θυμάστε ίσως 8 αντιδραστήρες ε, έκλεισαν ε, πριν από το προγραμματισμένο τέλος της ζωής τους για να ενταχθούν οι χώρες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αντάλλαγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να δώσει οικονομική βοήθεια στις τρεις ε, χώρες αυτές. Βλέπετε εδώ τις 8 διαφάνειες, 2 στην Ιγναλίνα, στη Λιθουανία, 2 ε, στο Μποχούνιτσε της Σλοβακίας και 4 ε, στο Κόσλο στη Βουλγαρία. Οπότε να σας πω πρώτα απ' όλα, βλέπετε και τις ημερομηνίε ε, όταν έκλεισαν. Η τελευταία η οποία έκλεισε ήταν η δεύτερη μονάδα της Ιγναλίνα που έκλεισε οριστικά το 2009. Πρώτη δηλώση που έχω να κάνω είναι ότι τώρα η αποσυναρμολόγηση έχει φτάσει πλέον σε στάδιο μη αναστρέψιμο και έχει προχωρήσει πάρα πολύ καλά στην τελευταία αυτή περίοδο που ξεκίνησε το 2014. Έχουμε επιτύχει τους περισσότερους στόχους και ο προγραμματισμός πηγαίνει κανονικά σύμφωνα με τις ε, ημερομηνίες που είχαμε υπολογίσει πριν. Αν δούμε το πρόγραμμα Ιγναλίνα, θεωρώ ότι αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι λόγω της ε, θέσεως ε, σε λειτουργία της ε, εγκατάστασης αποθήκευσης του εξαντλημένου καυσίμου. Μπορέσαμε να φέρουμε όλο το καύσιμο από τους οντερεστήρες στην εγκυναλίνα και όπως βλέπετε στις εικόνες έχουμε στην εικόνα που γράφει μετά έχουμε τα δοχεία με το καύσιμο και προχωράμε κανονικά και πάρα πολύ καλά και μπροστά από το πρόγραμμα μάλιστα. Πάλι για να σας δώσω πάλι μια ιδέα του τι συμβαίνει στο άλλο κομμάτι του περνικού εργοστασίου όπου βρίσκονται οι στρόβιλοι για να σας δώσω μια ιδέα του τι μιλάμε η αίθουσα των στροβίλων έχει μήκος 800 μέτρων Οπότε αρκετά μεγάλη οπότε ε, η αίθουσα των στροβίλων του εντελεστήρα 1 είναι βασικά άδεια το ίδιο και η δεύτερη αίθουσα και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων που συλλέγουν τα απόβλητα που μιλάμε για απόβλητα χαμηλού επίπεδου και θα επανέλθω σε αυτό όταν θα μιλήσουμε για τον Μπουχούνιτσε λειτουργεί και αυτή πλήρως. Λοιπόν, εάν δούμε το Κοσλοντούι τώρα στη Βουλγαρία, έχουμε τέσσερις αντιδραστήρες και εδώ πέρα επίσης είναι ενδιαφέρον το ότι όλος ο εξοπλισμός που περιέχεται έχει αποσυναρμολογηθεί πλήρως, μάλιστα έχουν επιτύχει αυτά τα ορόσημα τον Αύγουστο φέτος η λειτουργία αυτή τη στιγμή η επιχείρηση προχωράει προς την αποσυναρμολόγηση του εσωτερικού των αντιδραστήρων που είναι βεβαίως ε, το πιο λεπτό κομμάτι της διαδικασίας. Ε, δύο σημεία πρέπει να τονιστούν εδώ πέρα νομίζω. Το ένα είναι ότι το αποθετήριο των αποβλήτων που χρειάζεται για τα απόβλητα μεσαίου και υψηλού επίπεδου κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή βλέπετε την εικόνα εκεί στα αριστερά και ταυτόχρονα υπάρχει μια πειραματική εγκατάσταση το λεγόμενο όπλο πλάσματος ε, που χρησιμοποιείται για τη μείωση του όγκου των πυρηνικών αποβλήτων και είναι κάτι το οποίο βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εγκαταστάσεις. Ο τύπος ε, της ε, μείωσης του όγκου που μπορεί να επιτύχει μια τέτοια εγκατάσταση είναι της τάξεως του 20. Ε, λειτουργεί λοιπόν και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι όχι απλά συμβατό με το περιβάλλον αλλά και οικονομικά αποδοτικό στο πλαίσιο της συνολικής πάυσης λειτουργίας. Λοιπόν, εάν δούμε τώρα το τρίτο πρόγραμμα στο Μποχούνιτσε Έχουμε δύο αντιδραστήρες, ίδιου ε, τύπου με τους αντιδραστήρες του Κοσλοντούι. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει προχωρήσει πιο πολύ στην εφαρμογή του. Να σας δείξω αυτές τις εικόνες εδώ. Ε, βλέπετε πάλι και την αίθουσα των στροβίλων που είναι άδεια και βλέπετε επίσης ότι το τοπίο στον Μποχούνιτσε έχει αλλάξει αρκετά υπήρχαν ε, τέσσερις ε, πύργοι ψήξης ε, που σχετίζονταν με τους τέσσερις δραστηρίες. Λοιπόν, δύο αντιδραστήριες λειτουργούν ακόμα και οι τέσσερις πύργοι έχουν αποσυναρμολογηθεί πλήρως. Το πρόγραμμα αυτό, όπως είπα, έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο γιατί πράγματι ημερομηνία στόχος για την ολοκλήρωση είναι το 2025. Το εσωτερικό των αντιδραστήρων ήδη το έχουμε επεξεργαστεί. Βλέπετε πως ε, έχουμε την διαδικασία που αφορά το κύκλωμα του, το πρωτογενές κύκλωμα του εσωτερικού του αντιδραστήρα. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια τα οποία κόβονται και υπάρχει ε, χειρισμός τους ε, και μετά από την διαδικασία αυτή θα απελευθερωθούν. Σημαντικό είναι και αναφέρομαι εδώ σε ένα απλό παράδειγμα να αντιληφθούμε του τι προκύπτει ως απόβλητα από την διαδικασία πάυσης λειτουργίας όπως βλέπετε 90% των υλικών ε, μπορούν ε, μετά την διαδικασία αυτή να πάνε να ξαναχρησιμοποιηθούν ε, τα μέταλλα πάνε για σκράπ τσιμεντένιες δομές επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιαχτούν καινούργιοι δρόμοι 10% είναι απόβλητα χαμηλού και πολύ χαμηλού επίπεδου, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία πριν ε, ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία πάυσης λειτουργίας να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις εκείνες οι οποίες θα δεχτούν τέτοια απόβλητα. Οπότε όταν ακούτε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 90 κλειστοί πυρηνικοί δραστήρες, αλλά τρεις έχουν πλήρως από αποσυναρμολογηθεί. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι πράγματι ε, τα αποθετήρια των αποβλήτων. Το κομμάτι το οποίο απομένει είναι είτε εξαντλημένα καύσιμα είτε απόβλητα υψηλού επίπεδου για το οποίο απαιτείται μια βαθιά γεωλογική απόθεση. Αυτό προτιμούμε. Ε, καμία από τις τρεις ώρες. δεν έχουν τέτοια αποθετήρια. Η διαφάνεια επίσης σας δίνει μια εικόνα οπτική από πλευράς τόνων του πόσοι τόνοι υλικών προκύπτουν από την διαδικασία. Λοιπόν, να δούμε τώρα την χρηματοδότηση. Σας εξήγησα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μεγάλο μέρος του κόστους ε, που σχετίζεται με την διαδικασία. Βλέπετε στα αριστερά για τα τρία έργα τα κονδύλια τα οποία είναι δεσμευμένα μέχρι το τέλος του 2020 και στην επόμενη στήλη βλέπετε το προτινόμενο ποσό στο επόμενο πι πι από την Κομισιόν. Επίσης βλέπετε το ύψος ε, των συνσφορών και σε απόλυτες ε, τιμές και σε ποσοστό των τριών δικαιούχων χωρών όσον αφορά τους ε, στόχους ε, του επόμενου πι δελτα έχουμε ξεκάθαρα τον στόχο της ολοκλήρωσης ε, της παύσης λειτουργίας του Μποχούνιτσε το 2025 και του να προχωρήσει η υπόθεση με το Κόσλο Ντούι εντός του προπολογισμού που έχουμε προτείνει. Η Γναλίνα είναι τελείως διαφορετική. Είναι άλλος αντιδραστήρας με γραφίτι και η αποσυναρμολόγηση του πυρήνα αφού βγει το κάψιμο θα είναι η κυρία πρόκληση στο επόμενο πι δελτα πι θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τα εργαλεία, νομίζω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν σημαντικές συνέργειες μεταξύ των τριών προγραμμάτων. Υπάρχουν άμεσες συνέργειες μεταξύ του Μποχούνιτσε και του Κοσλοντούι, γιατί είναι ο ίδιος τύπος αντιδραστήρα, όπως είπα ήδη. Και η συνέργεια αυτή μπορεί να καταλήξει στο να υπάρχει ανταλλαγή πρακτικών, οπωσδήποτε, αλλά και στο να χρησιμοποιηθούν ξανά τα ίδια εργαλεία και μέσα. Ενώ για το ζήτημα της αποσυναρμολόγησης ε, του πυρήνα με γραφίτη στην Ιγναλίνα προσπαθούμε ακριβώς ε, να βρούμε την καλύτερη γνωμοσύνη που υπάρχει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια, επιλογή, μια μελέτη επιλογών και αναμένεται πως η σύμβαση για την αποσυναρμολόγηση του πυρήνα θα συναυθεί το 2022. Να πω επίσης πως υπάρχει μεγάλος αριθμός ε, κλεισίματος τέτοιων εγκαταστάσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιμένουν αποσυναρμολόγηση. Υπάρχει μια μεγάλη αγορά λοιπόν που αναμένεται να μεγαλώσει κι άλλο και έχει σημασία να αναλάβουν οι καλύτεροι και πιο καταρτισμένοι. Αυτά είναι λοιπόν τα δυνητικά και δευτερεύοντα ωφέλη που μπορούν να έχουν αυτά τα προγράμματα. Οπότε δεν είναι ε, μόνο η άμεση συναρμολόγηση και το ότι δεν θα υπάρχει πλέον ραδιολογικός κίνδυνος από τη λειτουργία των εργοστασίων αλλά και το ότι οι εταιρείες αυτές μπορούν πλέον να εξάγουν τεχνογνωσία σε άλλες χώρες. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στην διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Gariba. Ευχαριστούμε κύριε Γκαρίμπα. Παρακαλώ, έχετε ερωτήσεις ή σχόλια. Ο κύριος Γκάιερ πρώτος ζήτησε το λόγο ή όχι. Όχι, ο κύριος Χάιζελ μάλλον. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Καρύμπα για την ενημέρωση. Πολύ άρτια έκθεση και αμερόληπτη. Είναι σημαντικό να κάνουμε ανταλλαγή εμπειριών σε αυτή τη σημαντική διαδικασία παροπλισμού των πυρηνικών σταθμών και τα τρία κράτη-μέλη ακόμη και πριν ε, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκάστηκαν να δεσμευτούν ότι θα κλείσουν οριστικά τα πυρηνικά τους εργοστάσια και τους ε, παλιούς επιρχιωμένους τους αντιδραστήρες και το έκαναν, τήρησαν την υπόσχεσή τους. Και αυτό είναι σημαντικό και αναμενόμενο, γιατί είναι θέμα ασφάλειας πυρηνικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει ε, την αποσυναρμολόγηση και τον παροπλισμό αυτών των πυρηνικών ε, σταθμών. Ερωτώ, υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά κενά, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σλοβακίας, γιατί εγώ είμαι Σλοβάκος και διαρωτώ με αν υπάρχει κάποιο κενό χρηματοδοτικό. Και αν ε, πιστεύετε ότι στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το χρηματοδοτικό κενό ή θα, θα στηρίξουμε τις χώρες να το καλύψουν. Αν υπάρχει τέτοιο χρηματοδοτικό κενό, μήπως υπάρχει κίνδυνος να υποσκαφθεί ε, ο παροπλισμός ή να μην ολοκληρωθεί εγκαίρως, δηλαδή για τη Σλοβακία μέχρι το 2025 και για τη Βουλγαρία μέχρι το 2030. Μήπως καθυστερήσει ο παροπλισμός, η ολοκλήρωση του παροπλισμού λόγω χρηματοδοτικού κενού. Γιατί αυτή η περιπτώση ε, τι θα συμβουλεύατε τις σλοβακικές και βουλγαρικές αρχές προκειμένου να τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους εγκαίρως. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εγώ ε, εργάστηκα για χρόνια στην Ιγναλίνα, είναι η γενέτειρά μου. Ε, έζησα 30 χρόνια εκεί, τέλεσα και δήμαρχος της Ιγναλίνα και πολλά στοιχεία της πόλης αυτή συνδέονται με τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού. Γνωρίζω λοιπόν ε, ε, εκ των έσω την κατάσταση. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή μας που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, για το θέμα αυτό και υπερψήφισε το ψήφισμα του προηγούμενου κοινοβουλίου, της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας για το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λυπάμαι ιδιαίτερος που στα εισαγωγικά της σχόλια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι τους κανονισμούς και την για την επόμενη περίοδο 2020-2027 θα επιτρέψει τη Λιθουανία να ολοκληρώσει τον παροπλισμό ε, του πυρηνικού σταθμού και να αξιοποιήσει ε, το γραφίτι. Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί ε, τα ποσά που έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα, 260 εκατομμύρια, δεν αρκούν για την ε, επεξεργασία ή τη διάθεση του εξαντλημένου γραφίτη, του πυρήνα, του αντιδραστήρα. 780 εκατομμύρια χρειάζονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διάθεσης του χρησιμοποιημένου γραφίτη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζήτησε αύξηση της συγχρηματοδότησης από τη Λιθουανία και στη συνθήκη τίποτα δεν αναφέρεται για το συντελεστή χρηματοδότηση. Η Λιθουανία δεσμεύτηκε στο 14% χρηματοδότηση ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί 20% χρηματοδότηση από τη Λιθουανία. Και στην έκθεσή σας δεν μας αναφέρεται τίποτα για το θέμα αυτό. Τι γίνεται με τη διάθεση του εξαντλημένου καυσίμου που θα πρέπει να αποθηκευθεί σε κάποιους χώρους διάθεσης και μάλιστα κάψιμο που χρησιμοποιήθηκε πριν από 25 χρόνια πρέπει να ε, διατεθεί οριστικά γιατί μετά από 25 χρόνια δεν θα μπορούμε πια να μιλούμε για βιώσιμη αποθήκευση αναγκαστικά θα πρέπει να πάει σε χώρο ταφή, σε χώρο διάθεσης χωματερή. Στο παρελθόν όταν υπήρχε κίνδυνος ε, διαρροής ε, ραδιενέργειας ήταν πολύ σοβαρό. Υπάρχει πολλοί κόσμος όμως που εργάζεται σε περιβάλλον με χαμηλής ραδιενέργειας ή διαχειρίζεται υλικά που έχουν ε, μία μικρή ακτινοβολία. Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Δεν κινδυνεύει η υγεία των εργαζομένων εκεί. Γνωρίζει την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται να εκπονήσει μελέτες ή έρευνες σχετικά για να δούμε πόσο θα επηρεαστεί η ανθρώπινη γέη ή το περιβάλλον μετά από 20-25 χρόνια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια σταθερή έκθεση σε ραδιενεργό περιβάλλον εδώ και τόσα χρόνια. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και το Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί ο παραπολισμός του πυροενικού εργοστασίου ήταν προαπαιτούμενο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί στηρίσαμε την υποχρέωσή μα, κλείσαμε του αντιδραστήρε, τους αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει την περιοχή. Από το 2014 όμως και μετά ε, αθετεί την υπόσχεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η κατάσταση στην περιοχή της Ιγναλίνα επιδεινώθηκε. Μία πόλη ε, 34.000 κατοίκων έμεινε με ε, ελάχιστο πληθυσμό, με λιγότερους από τους μίσους, 18.000. Οπότε δεν θα πρέπει να συνεχίσετε και για την επόμενη περίοδο την ε, περιφερειακή στήριξη της Ιγναλίνα. Κυρία Πόλσον. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ πιο σύντομη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Έχω μια ερώτηση. Μιλήσατε για όπλο πλάσματος για τη μείωση του όγκου. Μάλιστα. Ε, αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό και θα ήθελα να, κάνω, να γνωρίζω αν αυτό το project θα έχει οικονομικά ωφέλη για την πυρηνική βιομηχανία, γιατί θα είναι εκατοντάδες οι σταθμοί παγκοσμίω που προχωρούν προς τον παροπλισμό τα επόμενα χρόνια. στην, ε, ε, μόλις εκδόθηκε η παγκόσμια έκθεση για την κατάσταση των πυρηνικών οπότε ο μέσος ε, σταθμός εκεί υπολογίζεται πως έχει διάρκεια ζωής 30 χρόνια οπότε τα κόστη είναι τεράστια, πολύ ε, εντυπωσιακά τα νούμερα και μόλις έμαθα από εσά ότι και άλλο κόστος μας περιμένει τα επόμενα χρόνια. Έχει κανείς υπολογίσει πώς ε, δαπανηρή θα ήταν η κιλοβατόρα αν τουλάχιστον είχε ε, υπολογιστεί και το κόστος παροπλισμού εξ αρχής. Ο Πομπάρ. Oui, merci pour euh, ce... Ε, σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Έχω τρία σύντομα ερωτήματα. Κάποια πράγματα έχουν ήδη υποθεί ίσως. Στην πρώτη, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι στη μελέτη αναφέρεται αντικειμενικά και στις ημερομηνίε για τον παραπλησμό τριών ε, πυρηνικών σταθμών. Όμως πρόκειται για τελείως νέο τεχνολογικό επίτευγμα. Εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε τεχνολογικές δυσκολίες ε, ή εμπόδια που ε, μπορεί να εμποδίσουν ε, τη δίδυση αυτών των ημερομηνιών, γιατί ξέρουμε ότι καθημερινά αντιμετωπίζονται νέες προκλήσεις. Έπειτα, το ερώτημα του συναδέλφου. Γνωρίζουμε ότι στον τομέα των πυρηνικών υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά τα εργοτάξια, τα οποία χρηματοδοτούμε εμείς τα προγράμματα παροπλισμού. Κατά πόσο αυτό η χρηματοδότηση συνοδεύεται με όρους και προδιαγραφές για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται εκεί, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως το πρόβλημα της πυρηνικής ραδιενέργειας είναι πολύ σημαντικά. Τρίτον, εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ξεπερασμένη και πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Το θέμα είναι όμως με βάση τον παροπλισμό αυτών των ε, αντιδραστήρων που είναι ένα συγκεκριμένο είδος μπορούμε να αποθηκεύσουμε τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον παροπλισμό άλλων πυρηνικών ε, ε, αντιδραστήρων δεύτερης και τρίτης γενεάς. Ευχαριστώ. Thank Και εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Αφόσον όχι, θα ε, ζητήσω από τον κύριο Γκαρίμπα να κλείσει. Ε, και να απαντήσει, απαντώντας μάλλον σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη σειρά των ερωτήσεων καθώς αυτές τέθηκαν. Όσον αφορά το ερώτημα του κύριου Άιζελ. Υπάρχουν όντως κενά. 19 εκατομμύρια ευρώ και όπως βλέπετε στην πρόταση της Κομισιόν έχουμε προτείνει 63 εκατομμύρια. Αν προσθέσουμε και το κανονικό ποσοστό που έχει συμβάλει μέχρι στιγμή η Σλοβακία θα καλυφθεί τελείως το κενό. Ε, όχι, δεν περιμένουμε λοιπόν να έχουμε κανένα πρόβλημα για την ολοκλήρωση του project αυτού το 2025 με τη βάση τις ε, δημοσιονομικές προβλέψεις που έχουμε σήμερα. τα ερωτήματα του κύριου Ροπέ ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι υπάρχει ε, διαφορά απόψεων ανάμεσα στην πρόταση της Κομισιόν και την έκθεση που ψήφισε το Κοινοβούλιο. Εκεί όπου δεν υπάρχει διαφορά απόψεων είναι για το ποσό που χρειάζεται για την επιχείρηση αυτή μέχρι το 2027. Και θα πρέπει να σας πω ότι τώρα είναι θέμα της Δημοσιονομικής Αρχής να αποφασίσει τελικά τι ποσό θα θελήσει να χορηγήσει ανάμεσα στο Συμβούλιο δηλαδή και Κοινοβούλιο στη συγκεκριμένη, ε, ε στο συγκεκριμένο project. Η, η Κομισιόν είναι σε διάλογο με τις λιθωνικές αρχές επ' αυτού. Και τώρα, όπως είπα, εξαρτάται τα δύο σκέλη της Δημοσιονομικής Αρχής να λάβουν την απόφαση. Ε, τώρα, μόνιμη αποθήκευση. Η ψηλά ραδιενεργών αποβλήτων είναι εκτός του πεδίου του προγράμματος αυτού και ανέκαθεν ήταν στις προτάσεις για το πρόγραμμα 2001-2027 δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο και μάλιστα αποκλείεται ρητά τα αποθετήρια αποβλήτων που δημιουργούνται στο στην Ιγναλίνα ε, έχουν σχεδιαστεί για μια διάρκεια ζωής 15 ετών. Είναι σημαντικό να τονίζουμε ότι ένας από τους δείκτες που έχουμε για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών είναι ο αριθμός των περιστατικών ή ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων για την ώρα σας πω ότι δεν έχουμε κανένα εργατικό ατύχημα. Και από το 2014 η Κομισιόν μετά από την υιοθέτηση των σχετικών κανονισμών του Συμβουλίου σταμάτησε να στηρίζει τα ενεργειακά προγράμματα που συνόδευαν τον παροπλισμό των πυρηνικών εργοστασίων αρχικά από το 2002 μέχρι και το 2013 διάφορα ενεργειακά προγράμματα είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποκαταστήσουν την έλλειψη παραγωγής ηλεκτρισμού που οφειλόταν στον παροπλισμό και το πρώιμο κλείσιμο του εργοστασίου και από την άλλη πλευρά την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις εν λόγω χώρες. Οπότε, τα project τα οποία χρηματοδοτήθηκαν πριν από το 2013 εξακολουθούν να κλείνουν στις τρεις χώρες αλλά οι κανονισμοί του Συμβουλίου δεν επιτρέπουν περαιτέρω χρηματοδότηση από τα κονδύλια παροπλισμού για αυτό το είδος τα προγράμματα. Αυτό που είναι όμως δυνατόν να γίνει, και αυτό εξαρτάται από τη βούληση των κρατών μελών, είναι να χρησιμοποιήσουν τα περιφερειακά ταμεία και τα ταμεία συνοχής για να στηρίξουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Τώρα, το όπλο πλάσματος, ναι, όντως ε, αφορά ε, υλικό χαμηλής ραδινέργειας, ε, αλλά ο βασικός στόχος είναι, αν δείτε τον μεγάλο όγκο αυτών των υλικών και το μεγάλο τονάζ, σημαίνει, όταν λειτουργεί σωστά, πως μικριώνει τις ανάγκες για χώρο και το κόστος της αποθήκευσης αν έχουμε υπολογίσει το κόστος του παραπλησμού στις κιλοβατόρα. Η Κομισιόν του 2017 δημοσίευσε ε, το ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο τακτικά δημοσιεύουμε, όπου περιλαμβάνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά το, τελευ... τέλος του κύκλου του καυσίμου και εκεί βλέπουμε όλες τις προβλέψεις των κρατών για το κόστος του παροπλισμού από τη μια, από το μια πλευρά και την τελική απόθεση των πυρηνικών αποβλήτων από την άλλη. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ξεχωριστά αν σας ενδιαφέρει. Η μέρα ολοκλήρωσης των προγραμμάτων, όπως είδατε, Έχουμε έναν αρκετά ευρύ ορίζοντα. Αυτό που είναι σημαντικό όμω να παρατηρήσουμε εδώ και θα ήθελα να το προσθέσω αυτό σε σχέση με την απάντηση που έδωσα για το σημείο που αφορούσε τη Λιθουανία. Ε, έχουμε λοιπόν το γεγονός ότι καλύπτουμε διάφορα πολιετή δημοσιονομικά προγράμματα. Ε, το σημαντικό όμως σημείο είναι ότι υπάρχει μια διαρκής πρόβλεψη χρημάτων, κονδυλίων μέχρι το τέλος ε, της ε, επιχείρησης παροπλισμού γιατί Σοβλαβακία είμαστε αρκετά βέβαιοι πως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία το 2025. Τώρα για την Βουλγαρία ήδη πάμε προς το 2030 οπότε εκεί θα άφηνα ένα μεγαλύτερο περιθώριο εκτίμησης και όπως ανέφερα για την Ιγκυναλίνα θα πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα σημαντικό στον παροπλισμό των πυρήνων γραφίτη. Αλλά αυτό ε, βάζουμε χρονικό όριο το 2030, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα πετύχει αυτή η, αυτό το εγχείρημα που είναι πρώτη φορά που γίνεται. Γι' αυτό δεν θα ήταν συνετό να δώσουμε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για αυτό το συγκεκριμένο σημείο για την Ιγναλίνα. Τώρα, τα κριτήρια για την ασφάλεια ορίζονται από δύο νομοθετήματα, τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας όσον αφορά την προστασία του εργαζομένου, νέα οδηγία του 2014 υπό τη συνθήκη Euratom, καθώς και η οδηγία πυρηνικής ασφάλειας που επιβάλλει συγκεκριμένες είδη αδειών που πρέπει να εκδοθούν από τις εθνικές αρχές και ούτω καθεξής. Πρόκειται δηλαδή εκεί αυτό, αυτά όλα παρακολουθούνται από την Επιτροπή που επαληθεύει το είδος του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν τα κρατημέλη για να ελέγχουν το επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων και της ραδιενέργειας του περιβάλλον. υπάρχουν δηλαδή διάφορα συνδυασμένα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ρωτήσατε επίσης Υπάρχει επίσης, ε, ρωτήσατε αν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης ε, το, για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που, που αποσυναρμολογούνται και είναι πρώτης γενεάς και σίγουρα στη δικό του σχεδιασμό δεν είχε κανείς σκεφτεί παροπλισμό. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική για τους αντιδραστήρες κυρίως του τρίτου, της τρίτης γενεάς όπου στο σχεδιασμό ήδη λαμβάνεται υπόψη ότι θα πρέπει να παροπλιστούν κάποτε. Δεύτερον, προσπαθούσα στην παρουσίασή μου να κάνω σαφή διάκριση ανάμεσα στους αντιδραστήρες με πυρήνα γραφητή όπως την Ιγναλίνα που ε, είναι ιδιαίτερη πρόκληση λόγω αυτού του γεγονότος και τους ε, αντιδραστήρες που ρυθμίζονται με το νερό και για τους οποίους δεν υπάρχει ιδιαίτερη τεχνολογική πρόκληση για την αποσυναρμολόγηση. Πρόκειται για βιομηχανική επιχείρηση Τα κανονικά λοιπόν εκεί ε, κομμάτια ε, δεν, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη πρόκληση και γι' αυτό στο Πογούνιζε επειδή έχει ε, το βασικό κύκλωμα, δηλαδή ο ίδιος αντιδραστήρας ε, ε, καθαριστεί, νομίζω πως θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρόνο διάγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Καρύμπα από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Σας ευχαριστώ και εσάς και αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη και έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνεδρίαση στην ώρα της. Επόμενη μας συνεδρίαση 17 Οκτωβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων. Σας ευχαριστώ όλους.